Ja, good afternoon. Ich κυρίες και ε, χαιρετώ για την ε, συνέχιση των εργασιών μας. Έχουμε, είχαμε αναβάλει ένα σημείο της ημερήσιας διάταξη, πρόκειται για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική και τη σχετική ρύθμιση. Ε, οι εισηγητές είναι ο Τάμας η Γιάννα Ιβάνοβα και κάποιοι άλλοι. Και από το ελεγκτικό συνέδριο καλωσορίζουμε τον κύριο Κρετά. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πρέπει να ακούσουμε αμέσως τον κύριο Κρετά ή επιθυμούν να πάρουν το λόγο οι εισηγητές. Όχι, ο κύριος ε, Κρετά θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, σημερινή πρόσκληση, ούτως ώστε να ε, γνωμοδοτήσει και το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή η πρόταση βασίζεται στα τέσσερα βασικά προγράμματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση και βασίστηκε στις διαπιστώσεις ε, του συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή της και στις επιμέρους ειδικέ εκθέσεις. Ε, τέσσερα είναι τα βασικά σημεία της παρουσίασής μου. Πρώτον, η απλούστευση της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ανταποκριθεί σε διάφορε παρατηρήσει ε, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ω προ την απλοποίηση του συστήματο. Θα πάρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτον, ε, το καθεστώς των βασικών πληρωμών θα αντικαταστήσει δύο προηγούμενα καθεστώτα, το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και το καθεστώς της στρεματικής ενίσχυσης που εφαρμοζόταν στις χώρες που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004. Θα αντικαταστήσει λοιπόν αυτά τα δύο καθεστώτα και ο καθεστώ, το καθεστώς ε, της ενιαίας ενίσχυσης με τις 20 διαφορετικές υποκατηγορίες θα εκλείψει. Οπότε ε, θα προκύψει σημαντική απλούστευση του συστήματος. Ένα άλλο παράδειγμα σχετίζεται με την θέσπιση ενός απλουστευμένου καθεστώτος για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ως προς άλλα σημεία αναγνώρισε τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως ε, κάνει προτάσεις που κατά τη γνώμη μας θα είναι δύσκολα εφαρμόσιμες ε, στην πράξη και θα επανέλθω σε αυτό εντός ολίγου. Γι' αυτό το λόγο συνολικά πιστεύει το Ελληνικό Συνέδριο ότι η κοινή γεωρική πολιτική εξακολουθεί να συνιστά ένα περίπλοκο ε, νομοθετικό σύνολο. Θα δώσω τρία συγκεκριμένα παραδείγματα που είναι χαρακτηριστικά ως προς την περιπλοκότητα του συστήματος. Ε, ας πάρουμε πρώτα την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το προτινόμενο πλαίσιο διατηρεί έξι διαφορετικά ε, κανονιστικά επίπεδα, ε, αρχίζοντας από τον κοινό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία μέχρι τις νομοθετικές διατάξεις εθνικό επίπεδο. Δεύτερο παράδειγμα σε σχέση με την ε, πολλαπλή συμμόρφωση. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου της πολλαπλής συμμόρφωσης οδηγώντας σε απλούστευση πλην όμως ε, μόνο κατ' επίφαση. Δηλαδή ε, ενοποιήσαμε σε ένα καθεστώς διάφορα διασκορπισμένα στο παρελθόν μέτρα αλλά δεν προκύπτει κατά τη γνώμη μας ουσιαστική απλοποίηση. Τρίτο παράδειγμα το θέμα των ενεργών γεωργών και του ανωτάτου του ορίου των ενισχύσεων. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε να είναι καλύτερα στοχευμένες οι ενισχύσεις προς τους ενεργούς γεωργούς και επίσης να προσδιορίσει ένα ανώτατο όριο για τις ενισχύσεις. Επ' αυτού θα συμφωνήσουμε με τη διάγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, ε, τα νομοθετικά μέτρα στη λεπτομέρεια τους φαίνονται υπερβολικά ε, περίπλοκα και κατά τη γνώμη μας ε, δύσκολα εφαρμόσιμα, τουλάχιστον όχι με αποτελεσματικό τρόπο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο γενικός κανονισμός θα μπορούσε να περιοριστεί σε έναν γενικό ορισμό του ενεργού γεωργού και να αφήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διακριτική ευχαίρεια να διαχειριστεί στην πράξη το νέο καθεστώς ε, ούτω ώστε να ανταποκριθεί ε, στις ε, πολλαπλές επιμέρους περιπτώσει που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή διότι δεν είναι κατά τη γνώμη μα πολύ αληθοφανέ εκ των προτέρων να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε όλες τι δυνατότητε που θα ανακύψουν στην πράξη μέσα σε ένα γενικό κείμενο νομοθετικού περιεχομένου Δεύτερον, ο στόχος ε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι σημαντικό αυτό το σημείο και θεωρούμε ότι οι νομοθετικές ε, προτάσεις δεν προσφέρουν επαρκώς σαφή απάντηση σχετικά με ε, τον στόχο των ενισχύσεων ε, που ε, χορηγούνται στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής. Οι προτάσεις που γίνονται εξακολουθούν να βασίζονται στους πόρους, στα μέσα της κοινή γεωρικής πολιτικής, δηλαδή στα κονδύλια που διοχετεύονται για την ε, χορήγηση διαφόρων ενισχύσεων και ως προς τα επιλέξιμα δικαιώματα. Αντί να εξετάζουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που όμως προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός, ε, ούτε προβλέπεται επαρκής ε, αποτίμηση των μέτρων αυτών. Τώρα, το να περάσουμε από την πολιτική των μέσων προς μια πολιτική αποτελεσμάτων ήταν ένας στόχος που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται πλήρω με τη συγκεκριμένη πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή και θα σα το αποδείξω με τέσσερα διαφορετικά παραδείγματα. Για τις άμεσες ενισχύσεις, αυτό είναι το πρώτο μου παράδειγμα, διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο δεν υπάρχει καμία μία ω προ το στόχο αυτόν στα αντίστοιχα άρθρα του διατακτικού του κανονισμού ούτε και ω προ τα αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής δεν αναφέρεται τίποτα. Δεύτερο παράδειγμα σε σχέση με την κατανομή των ενισχύσεων ε, στους δικαιούχου. Ε, ούτε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στον κανονισμό. Η κατανομή των ενισχύσεων ε, παραμένει λοιπόν όπως και σήμερα ε, το αποτέλεσμα μέτρηση σε βάση το, της έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης. Οι, μικρές, λοιπόν, εκμεταλ Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις λοιπόν θα λαμβάνουν την πλειοψηφία των ενισχύσεων. Τι γίνεται τώρα με τις ε, λιγότερο ευνοημένες ε, περιοχές, τι γίνεται με τους νέους ε, γεωργούς, θα δικαιούνται προς αύξηση ανά εκτάριο, αυτό έχει προβλεφθεί, όμως παρά, παρόλα αυτά τα θετικά βήματα θεωρούμε ότι υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή η εσωτερική αντίφαση υπήρχε και στην προηγούμενη ΚΑΠ ε, έγκυται αυτή η αντίφαση αφενός το ότι θέλουμε να στηρίξουμε το ατομικό εισόδημα ενώ δεν προσαρμόζουμε αυτό το ατομικό εισόδημα στις συγκεκριμένες περιστάσεις που διέπουν κάθε εκμετάλλευση. Δεν λαμβάνουμε υπόψη παραδείγματο χάρη το διαφορετικό κόστος που καλούνται να φέρουν οι γεωργοί ούτως ώστε να παράγουν ε, αυτά τα δημόσια αγαθά που περιμένει ο καταναλωτής από αυτούς. Τελευταίο παράδειγμα, σε σχέση με το στόχο της μεταρρύθμισης, πρόκειται για την ε, πολλαπλή συμμόρφωση και την ε, οικολογική διάσταση ε, που εισαγάγεται πλέον σε αυτό το καθεστώς των βασικών πληρωμών. Λοιπόν, ο στόχος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πολλαπλής συμμόρφωσης καθώς και της οικολογικής διάστασης ως προς τις άμεσες ενισχύσεις δεν προσδιορίζονται επαρκώ μέσα στην πρόταση. Κατά αυτόν τον τρόπο και επίσης συνειδητοποιούμε μάλλον ότι υπάρχουν μελέτε που αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων, όπω παραδείγματος χάρη ο προσδιορισμό των ζωνών οικολογικού ενδιαφέροντος, ε, τα τέτοια πορίσματα λαμβάνουν, ε, λαμβάνονται υπόψη αλλά όχι επαρκώς. Η βιοπικιλότητα τώρα. Υπάρχουν ε, άφθονα επιστημονικά στοιχεία για να δικαιολογηθεί η πρόταση κανονισμού, όμως δεν προσδιορίζονται οι στόχοι επαρκώς μέσα στον κανονισμό, ούτε και αναφέρονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή των μέτρων. Τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα, η ανάπτυξη της υπαίθρου. Στον τομέα αυτό το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει μία σειρά ε, στόχων και προτεραιοτήτων ε, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους. Παρά είναι διαφορετική, παρά είναι πολυάριθμοι στόχοι και οι προτεραιότητες ε, και κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι καλύτερα εστιασμένα τα μέτρα που προτείνουμε και λιγότερο περίπλοκα. Φτάνω στο τρίτο σημείο της μου η εποπτεία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την ε, θέσπιση συστημάτων διαχείριση και ελέγχου ε, σε εθνικό επίπεδο μετά τη θέση εφαρμογή τη μεταρρυθμισμένη κοινή γεωργική πολιτική. Οι οργανισμοί πληρωμή και οι οργανισμοί πιστοποίηση συγκεκριμένα. Θα κάνω δύο παρατηρήσει. Το κράτο μέλο εγκρίνει τι αρχέ πληρωμέ. Είναι οι αρχέ, οι φορεί που καταβάλουν στου δικαιούχου τι ενισχύσει. Είναι εθνικοί φορεί. Θεωρείται το ελεγκτικό συνέδριο πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι, ε, φέρει την ε, τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού θα πρέπει να εποπτεύει την συγκρότηση αυτών των εθνικών φορέων εξ αρχής ούτως ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτοί οι εθνικοί φορεί πληρωμής ώστε στη συνέχεια να αποφύγουμε μία σειρά από δυσκολίες που θα ανακύψουν συν το χρόνο. Ως προς ε, τους οργανισμούς επιστοποίησης τώρα. Δεν ε, λαμβάνουν την έγκριση από τα κράτη-μέλη, διορίζονται τα μέλη τους από τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί ως πηγή εγγύσεων το έργο αυτών των φορέων διαχείρισης. Γι' αυτό το λόγο Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έπρεπε να αναλάβει ένα ρόλο επαλήθευσης αυτών των συστημάτων, των συστημάτων δηλαδή που εφαρμόζουν οι εθνικοί φορεί πιστοποίησης, ούτως ώστε να επαληθεύεται, να ελέγχεται ε, η απόδοσή τους. Ένα δεύτερο σημείο που πάλι σχετίζεται με αυτούς τους φορείς πιστοποίησης είναι το εξής. προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεύρυνση του ρόλου αυτών των φορέων, ώστε να πιστοποιούν την νομιμότητα των πληρωμών. Όπως ξέρετε, σήμερα αυτοί οι φορείς έχουν μια περιορισμένη ευθύνη και ε, εξετάζουν την αξιοπιστία των λογαριασμών. Εδώ ο κανονισμός προτείνει επέκταση του ρόλου τους για να αναλάβουν και την πιστοποίηση της νομιμότητας των πληρωμών. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι πολύ χρήσιμο και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους. Όμως παρατηρήστε ε, την διατύπωση μέσα στον κανονισμό αυτής της πρόθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας εκπλήσει. Συγκεκριμένα, μελλοντικά προβλέπει ο κανονισμό ότι αυτοί οι φορεί πιστοποίηση θα εκδίδουν γνωμοδότηση όχι επί των λογαριασμών, αλλά επί των, της δήλωσης αξιοπιστίας ε, ε, της ε, διαχείρισης αυτών των φορέων, δηλαδή της δήλωσης που υπογράφει ο διευθυντής του διαχειριστικού φορέα. Κατά γνώμη όμως υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο να εκδώσει κάποιος γνωμοδότηση σε σχέση με τη διαχείριση και άλλο να πιστοποιείται έτσι με αυτή τη δήλωση η νομιμότητα των λογαριασμών. Αναρωτιόμαστε ακριβώς ποια είναι η έννοια ε, της ε, διατύπωσης αυτού του συγκεκριμένου άρθρου του Γενικού Κανονισμού. Περνάω στο τέταρτο και τελευταίο σημείο της παρουσίασής μου, αλλά θα πω πολλά, σας το λέω εξ αρχής. Εκαθάριση λογαριασμών και το θέμα της ε, μείωσης των πληρωμών σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια για να γίνει εκταμίευση. Πρώτα, εκαθάριση λογαριασμών. Για ε, το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι η διαδικασία καθάρισης λογαριασμών εξακολουθεί να αποκλίνει από το στόχο και από τον ορισμό της διαδικασίας αυτής σε δυνάμει του ε, κείμενου δημοσιονομικού κανονισμού άρθρου 53 και ως προς ε, τις εκτελεστικές διατάξεις του ίδιου κανονισμού άρθρου 42 των εφαρμοστικών διατάξεων. Υπενθύμιζε επανειλημμένα το ελεγκτικό συνέδριο ότι ο γενικό στόχο τη εκαθάριση των λογαριασμών συνίσταται στο να έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την τελική τη ευθύνη προ την εκτέλεση του προπολογισμού και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των γεωργικών δαπανών που εκτελούνται από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της συνδιαχείρισης. Για να αναλάβει αυτή την τελική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρώτον να προσδιορίσει το ύψος των δαπανών ε, που μπορούν να αποδοθούν στον προπολογισμό της Ένωσης γιατί έχουν πάγιο χαρακτήρα και αφιτέρουν να ε, απομακρύνει τις ε, παράτυπες δαπάνες. Όσε ε, τέτοιες πληρωμές είναι νομότυπε και μπορούν να αποδοθούν στον προπολογισμό υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ο προσδιορισμό του τελικού ποσού δεν ε, προβλέπεται μέσα σε αυτόν τον κανονισμό ω ευθύνη τη ευρωπαϊκή επιτροπή. Αυτό το ετήσιο συνολικό ποσό των δαπανών που βαρύνουν τον προπολογισμό της Ένωσης ε, δεν ε, προσδιορίζεται με θετικού χαρακτήρα απόφαση. Πάλι για την εκαθάριση των λογαριασμών διαπιστώνει το ελεγκτικό συνεδρίο ότι καμία ε, προτινόμενη τροποποίηση δεν διορθώνει το πρόβλημα των καταποκοπήν δημοσιονομικών διορθώσεων, εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε αναλύσει από διάφορες οπτικές ε, γωνίες ε, το εύρος χρήσης αυτού, του συστήματος των καταποκοπήν δημοσιονομικών διορθώσεων και ε, ε, αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι ε, το ποσό που προβλέπεται για τις δημοσιονομικές διορθώσεις διαφέρει από το ποσό που προβλέπεται για το ΕΤΠΑ, για το ΕΚΤ και για το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια των διαρθρωτικών ε, ταμείων, όταν προτείνει κατά αποκοπήν διόρθωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι το ύψος της παρατυπίας είναι χαμηλότερο ε, από την ε, κατά αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δυνατότητα να ε, ε, αποδείξουν ότι είναι υπερβολική δημοσιονομική διόρθωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπεται στο αντίστοιχο κομμάτι του κανονισμού σε σχέση με τις γεωργικές δαπάνες. Κάτι άλλο τώρα σε σχέση με τη μείωση των ε, ενισχύσεων. Ε, μείωση της ενίσχυσης ε, που μπορεί να ζητήσει ένας δικαιούχος ε, προβλέπεται από τον κανονισμό όταν κάποιοι όροι, κάποιες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο δικαιούχος δεν γίνονται σεβαστές. Το σχέδιο κανονισμού, και εδώ μιλάω συγκεκριμένα για το άρθρο 65, είναι ιδιαίτερα συγκεχημένο. εισαγάγει μία στη διαφοροποίηση εγώ τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η έννοια τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην μείωση των πληρωμών αφενό και αφετέρου των κυρώσεων υπομορφή μείωση ενισχύσεων. δεν διευκρινίζεται περαιτέρω αυτή η διαφοροποίηση. αν τώρα κάνουμε ένα άλμα και φτάσουμε στο άρθρο 97, ε, συνειδητοποιούμε ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι αυτές οι κυρώσεις υπό τη μορφή μειωμένων πληρωμών δεν έχουν επίπτωση επί της νομιμότητας των πληρωμών. Πάλι ξαφνιαζόμαστε με αυτή την διάταξη, διότι τι σημαίνει αυτό στην πράξη. ένα δικαιούχο που παραβιάζει τις κανονιστικές ε, διατάξεις ε, θα θεωρηθεί ως ε, ε, δικαιούχος ολόκληρης της ενίσχυσης θα θεωρείται απολύτως ε, νόμιμη πληρωμή, όμως θα υποχρεούται ο δικαιούχος να επιστρέψει λόγω της παρατυπίας ένα κομμάτι της πληρωμής υπό μορφή κύρωσης. Ποια πιο το νόημα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η διάταξη. Η μείωση ε, των ε, ενισχύσεων είναι ε, αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής της πολλαπλής συμμόρφωσης. Μέσω της μείωσης των ενισχύσεων επιδιώκουμε να επιφέρουμε μια, καλύτερη συμμόρφωση, αν θέλετε, με την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης. Δύο παρατηρήσεις από αυτού. Όταν μιλάμε για τη μείωση λόγω παραβιάσεων υποχρεώσεων ω προ την πολλαπλή συμμόρφωση, το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι πρόκειται εδώ για νομικέ υποχρεώσει όπω και όλε οι υπόλοιπε και ε, οι διαχειριστέ μονάδων εκμετάλλευση πρέπει να συμμορφωθούν σε αυτό τόσο ώστε να λάβουν στο ακέραιο τι ενισχύσει. Οποιαδήποτε παραβίαση των σχετικών διατάξεων καθιστά παράτυπη και παράνομη ε, την πληρωμή, κατά τη γνώμη μα. Δυστυχώ όμω δεν υιοθετεί τη διαστάση μέσα στον κανονισμό. Τέλος και πάλι για το ίδιο θέμα. Ε, διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο ότι το σύστημα μείωσης ε, των ε, πληρωμών λόγω της παραβίασης των υποχρεώσεων του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης αποδυναμώνεται με τη νέα πρόταση διότι το συνολικό ποσοστό μείωσης που προβλέπεται στον προηγούμενο κανονισμό ήταν περίπου στο 3%. Δεν υπάρχει όμως πλέον αυτό το ποσοστό στο νέο, στη νέα πρόταση κανονισμού. Θα σταματήσω εδώ. Α, όχι, να πω και κάτι άλλο κλείνοντας. Μην ξεχνάτε ότι η μεταρρύθμιση αυτή, μάλλον η υλοποίηση αυτή, ε, συνεπάγεται διοικητικό κόστος ε, κυρίως ε, για τα κράτη-μέλη που μπορεί να ανέλθει και στο 15% ως προς την διαχείριση των άμεσων πληρωμών. Θεωρεί το ελεγκτικό συνέδριο δεν υπήρξε επαρκή ενημέρωση που να καταδεικνύει ότι αυτό το επιπρόσθετο κόστος θα αντισταθμιστεί από ένα ε, θα αντισταθμιστεί από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και πρόεδρε δεν θέλω να κλείσω προτού τονίσω ε, πόσο χρήσιμε είναι οι επαφέ που είχαμε με του ε, εισηγητέ σα τους εισηγητές της Επιτροπής σας. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία μας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να κλείσω. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέτα ε, πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η παρουσίαση αυτή σε σχέση με ένα σημαντικότατο τομέα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς θα υπάρξουν κάποια ερωτήματα. Εγώ θεωρώ το αποτέλεσμα της έκθεσής σας πραγματικά να οδηγεί στο αίτημα μιας, ε, στο αίτημα του να πάυσει άμεσα μια τέτοιου είδους ε, μεταρρύθμιση. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τον εισηγητή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβέστερα ποια είναι τα αίτια για αυτή την αύξηση του γραφειοκρατικού κόστους και πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να την εμποδίσουμε. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής ε, τους εισηγητές ποιος επιθυμεί να πάρει το λόγο. Η κυρία Ιβάνοβα ή ο κύριος Ντόιτς. Δεν βλέπω την κυρία Χολμάιρ. Ε, Διαδικαστικό. Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια αντίδραση από τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν ξεκινήσουμε με τις δικές μας αντιδράσεις. Πρόεδρος, αν συμφωνεί η Επιτροπή, συνήθως ο κανόνας είναι ότι οι συγητές παίρνουν το λόγο. Όμω είναι πολύ σημαντικό σημείο και αν συμφωνεί η Επιτροπή μπορούμε να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εκπρόσωπο αυτής να προβεί σε δήλωση. Καλώ. συμφωνούν άπαντε. οι δύο συζητητές. Βλέπω ότι συμφωνούν. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει την ευγένεια να μας πει ποιος είναι σε θέση να απαντήσει. Ο κ. Πατσέκο, καλά το προφέρω το όνομα. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που μας δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε αμέσως μετά το αξιότιμο μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Κρετά, το οποίο χαιρετίζω και θα ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την γνωμοδότησή του, διότι πράγματι πρόκειται περί χρησιμοτά τη συνεισφορά τη εργασία μα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ Επίσης, μάλλον εκφράζω την ευαρέσκειά μου, ότι αναγνωρίζει το ελεκτικό συνέδριο τη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έλαβε υπόψη πολλές από τι συστάσεις, Κυρίω απλούστευση. Θα ήθελα να επισημάνω, όπως ανέφερε ο κύριος Χετάν εξάλλου, ότι όσον αφορά τον τύπο πληρωμών, συγχωνεύσαμε δύο μοντέλα ή όσον αφορά την εισαγωγή ενός απλουστευμένου ε, σύστημα για τους γεωργούς που ωφελεί όλους τους γεωργούς και στις χώρες που έχουν πιο μικρή διοικητική δυνατότητα ε, καλύπτει τα δύο τρίτα των γεωργών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την έννοια του ενεργού γεωργού το οποίο επεσήμανε και ο Σκρατέν ότι πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση που ζητά το ελεκτικό συνέδριο, αλλά πόρο απέχουμε από την απλούστευση που μπορούμε να επιφέρουμε. Θέλω να πω ότι σκεφτόμαστε, προβληματιζόμαστε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ορισμό του ενεργού γεωργού, ούτω ώστε οι ενεργοί γεωργοί και μόνο οι ενεργοί θα παίρνουν πληρωμές. Και δεν θέλουμε ορισμός να δημιουργήσει διοικητικό άκθο συμπληρωματικό για τα κρατη Και προβληματιζόμεθα, λέγω, επί αρνητικής που θα μπορούσε να ε, φροντίσει να πετύχουν το στόχο μας. Επίσης, αν θέσουμε και ένα όριο, ένα κάπινγκ, ανώτατο όριο, όσον αφορά την πιο ισότιμη κατανομή των ενισχύσεων των άμεσων. Όσον αφορά το σημαντικότερο ρόλο που δίνεται στους φορείς επιστοποίησης, που το χαιρετίζει αυτό και το ελεκτικό συνέδριο, θα δίνουν αμέσως μια δήλωση ε, όσον αφορά αξιοπιστία, όσον αφορά και τις οργανισμούς που κάνουν πληρωμές και την αξιοπιστία και τον τακτικό χαρακτήρα των συναλλαγών. Και σχετικά με αυτό θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ελέγχει τους οργανισμούς πιστοποίησης μέσω αναλύσεως κινδύνου, κάτι που συνέστησε και το ελεκτικό συνέδριο άλλωστε. Καλώς! Υπογραμμίζει στο Ελεκτικό Συνέδριο όμω η μεταρρύθμιση δεν είναι αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά την απλούστευση. Εδώ ήδη αναφέρθηκα στο θέμα, στην περίπτωση των ενεργών γεωργών, όπου εκεί θεωρούμε ότι είναι βάσιμη η κριτική που γίνεται και προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικέ ε, λύσει, όπω προανέφερα. Υπάρχει και η περίπτωση τύξω της υπαίθρου όπου το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι έχουμε πολλέ διοικητικέ πολλές και κανόνε ερεσιμότητας πολύ περίπλοκου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όσον αφορά την ανάπτυξη πέθρου, το στατικικό πλαίσιο, το κοινό που εφαρμόζεται σε όλα τα διθετικά ταμεία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου έχει ακριβώς σαν στόχο να εισαγάγει ένα συνεπές, συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο. Τι ούτω τρόπος θέλουμε να βρούμε απάντηση. Όσον αφορά την οικολογική πολλαπλή συμμόρφωση, θεωρούμε ότι η πρότασή μας ήδη περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των απαιτήσεων που υπήρχαν προηγουμένως. Εδώ, όπως και σε όλες τις πολιτικές, μέρημνά μας είναι απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και του κανονιστικού και να συμβάλλουμε στην εξυπηρέτηση των στόχων όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, τη βιοπικιλομορφία, την πολιτική των υδάτων, την υγεία ή την ευημερία των ζώων. Έχουμε πολλαπλούς στόχους, προφανώς θα κάνουμε απλούστευση, αλλά περιοριζόμαστε βέβαια εν αυτή τη ενία από τον επιδιωκόμενο στόχο. στόχο συγγνώμη. Ο κύριος Κρετά ήδη έδωσε κάποιο παράδειγμα ότι δεν ελέγχουμε ε, παρκώς τις άμεσες πληρωμές μας για ειδικές περιπτώσεις ή για συγκεκριμένες δαπάνες. Το κάνουμε στην περίπτωση αναπτύξεως υπαίθρου όπου εξετάζουμε ακριβώς ε, ποιο κέρδος υπάρχει, για, ποια είναι η απώλεια του κάθε γεωργού μάλλον για να πετύχουμε κάποιους στόχους Ποια είναι η διαφορά, αλλά στην περίπτωση των άμεσων πληρωμών, αν είχαμε να καθορίσουμε για κάθε γεωργό ποιο ήταν το ειδικό κόστος το οποίο θα πρέπει να αποζημιωθεί, θα αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση που θεωρούμε ότι θα αντέβαινε την πολιτική της απλούστευσης. Και θέλουμε εδώ ε, να ε, το αποφύγουμε. Λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι θα πρέπει να ελέγξουμε τις δαπάνες και ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή η αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και τη συνέπεια. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά λοιπόν η πρότασή μας ε, κάνει μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πράγματι, έχουμε σε άθρο το 110 πρόταση σχετική που αφορά τους οριζόντιους κανονισμούς που προβλέπει ρητά εκεί τη δημιουργία ενός πλαίσιου παρακολούθησης και αξιολόγησης για να προσμετρήσει τις επιδόσεις όλων των αγροτικών πολιτικών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Και έχουμε αναπτύξει και δείκτες και κάθε τέσσερα χρόνια ε, υποβάλλουμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτού του πλαισίου αξιολογήσεως και παρακολουθήσεως. Ε, όσον αφορά αυτά που είπε το Ελεκτικό Συνέδριο, την ανάγκη να δίνουμε στους οργανισμούς πληρωμής των κρατών μελών τον αναγκαίο χρόνο για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να προσαρμόσουν τα συστήματα και τι διαδικασίε του στι νέε αγροτικέ πολιτικέ, στην αγροτική πολιτική. Εκεί συμμεριζόμαστε απόλυτα, πλήρω αυτή την ανησυχία. Έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τους οργανισμούς πληρωμών και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστούν. Όμω, και σα επιστούμε εδώ την προσοχή, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι θα πρέπει οι αποφάσει να αφορά τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική να λαμβάνονται έγκαιρα και να δίνεται επαρκή χρόνο, ούτω ώστε πριν να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγέ, οι οργανισμοί πληρωμών και οι εθνικέ διοικήσει σε άλλου τομεί να μπορούν να είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να κάνουν τα δέοντα. Λοιπόν, σχόλια. Σχολείο τελικό από την πλευρά μου. Να υπενθυμίσω ότι η απλούστευση είναι σημαντικότατη αποτελεί για μας θεμελιώδες στοιχείο, όμως δεν είναι αυτός σκοπός. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να συγκρίσει με τους στόχους της πολιτικής μας όπως είναι η άμεση υποστήριξη, ε, μια πιο πράσινη γεωργία και καλή χρηματοπιστωτική διαχείριση. Πιστεύουμε ότι γέννη έχουμε πετύχει καλή ισορροπία, αλλά είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου προσεκτικότατα, μόλις τη λάβαμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της απλούστευσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ομοδότηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το ρόλο στους συγητές, καταρχήν στην κυρία Ιβάνοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρώτη της ε, παρέμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο, ιδιαίτερα τον κύριο Κρετάν για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για την ιδιαίτερα προσεκτική ανάλυση που μας κάνατε. Εγώ είμαι συγγήτρια για τη γνωμοδότηση όσον αφορά τον οριζόντιο κανονισμό θα σχολιάσω λοιπόν εν συντομία τη γνωμοδότηση από αυτή την ε, σκοπιά. Πιστεύω ότι ο κανονισμό αυτό χρειάζεται βελτιώσει όσον αφορά τα αποτελέσματα, την πρόληψη, την απλούστευση και την ανάλυση κόστου και ωφέλεια. Πρώτον, όσον αφορά τα αποτελέσματα, υποστηρίζω την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου ότι θα πρέπει να είναι ο κανονισμό προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και δεν υπάρχουν επαρκείς ε, προβλέψεις για μια χρηστή οικονομική διαχείριση. Χαίρομαι που άκουσα από την Επιτροπή ότι έχουν αναπτυχθεί κάποιοι δείκτες αποδοτικότητας και ελπίζουμε πραγματικά να τους δούμε να λειτουργούν και να καταμετρούν αποτελεσματικά την, ε, τα αποτελέσματα, ε, την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος. Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης, πιστεύω ότι είναι πάντοτε πιο φτηνό το να προλαμβάνει κανείς από το να επιδιορθώνει, να παρεμβαίνει σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Ε, θα πρέπει να ενισχυθούν λοιπόν τα μέτρα πρόληψης όσον αφορά τους φορείς, τους οργανισμούς πιστοποίησης και πληρωμών. Ε, θα πρέπει να μην γίνεται μία εκ των υστέρων ανάλυση Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση κόστους ωφέλειας ε, των νέων διατάξεων της πρότασης, ε, η αύξηση είναι στάξη του 50% ως εκτίμηση του κόστους των οργανισμών. Αλλά διαθέτουμε μια ανάλυση κόστους ωφέλειας, δηλαδή ποιες είναι ακριβώς οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα ωφέλη ε, θα είναι κατά 50% υψηλότερα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέταρτον, όσον αφορά την απλούστευση σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος ε, Κρετάν στην παρουσίασή του, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη απλούστευση στις διαδικασίες και θα ήθελα να γνωρίσω τις προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πρότασης αλλά παραμένουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την διασταυρούμενη συμμόρφωση ε, και υπάρχουν διάφορα επίπεδα λήψη αποφάσεων. Τώρα έχω κάποια ερωτήματα προς την Επιτροπή που να μεν ε, τέθηκαν τον κύριο Κρετάν. Δεν άκουσα τις απαντήσεις, γι' αυτό θα επιτρέψατε μου να τα επαναλάβω. Πρώτον, όσον αφορά τους οργανισμούς πιστοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ε, γνωμοδότησης ή μάλλον του κανονισμού τα, οι οργανισμοί πιστοποίησης ε, θα αποφαίνονται όσον αφορά την δήλωση αξιοπιστίας και όχι τους ίδιους τους λογαριασμούς θα αξιολογούν λοιπόν την ίδια τη αξιοπιστία και όχι την ε, δήλωση αυτή καθ' αυτή. Ε, Διερωτώ ποιο είναι ο λόγο αλλαγή, αν το κατανοήσαμε καλά και αν μπορείτε να μα το εξηγήσετε. Θεωρείτε ότι αυτή η διαδικασία θα μα δώσει μια υγιή βάση για τη διενέργεια ελέγχου και για την παρακολούθηση. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση σε σχέση με την καθάριση των λογαριασμών. Διερωτώ με γιατί στο πεδίο της γεωργική πολιτικής δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μοντέλο όπως είναι στα διαρθρωτικά ταμεία όπου μπορούμε να έχουμε πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τις ε, ατασταλίες, για τις παρατυπίες ε, παρά για την διόρθωση των σφαλμάτων. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο θέμα, θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι ακριβώς η έννοια που προσδίδεται στο, στις κυρώσεις. Ιδιαίτερα στο άρθρο 97 που επιδέχεται πολλά περιθώρια ερμηνείας. Δηλαδή τα πρόστιμα δεν μπορούν ε, να καταμετρηθούν επακριβώς σε σχέση με τα αξιολογούμενα σφάλματα. Μπορείτε, να μας διευκρινίσετε. Τώρα όσον αφορά τη διασταυρώμενη συμμόρφωση ε, αναφέρθηκε ότι στην πρόταση της Επιτροπής, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, περισσότεροι γεωργοί θα αποκλειστούν από αυτή τη διαδικασία. Αλλά σήμερα έχουμε ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης που καταλαμβάνονται μόνο από μικρές ε, καλλιέργειες, από μικρούς καλλιεργητές. Όλες αυτές οι περιοχές πρόκειται να εξαιρεθούν από αυτούς τους κανονισμούς, τους κανόνες. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτή η έλεγχη είναι ιδιαιτέρως ε, πολύπλοκη και ε, χρονοβόρη. Αλλά ποια είναι ακριβώς ε, η γνώμη σας. Θέλετε να γίνει μια ad hoc δειγματοληψία ή θα πρέπει να εγκαταλειφθούν πλήρως αυτοί οι έλεγχοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνεγητής Κύριος Τόμας Ντόιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εφόσον μου το επιτρέπετε, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις γενικής φύσεως καταρχήν και στη συνέχεια θα επισέλθω σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τον κύριο Κρετέ, καθώς ε, το, επειδή το ελεγκτικό συνέδριο πραγματικά έκανε μια πολύ καλή έκθεση. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους γιατί πραγματικά πρόκειται για μια υποδειγματική συνεργασία με τον κύριο Κρετά. Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και τα προηγούμενα χρόνια τα προηγούμενα χρόνια η κοινή γεωργική πολιτική ήταν ένας μεγάλος τομέας και αυτό θα πρόκειται να αλλάξει για το χρονικό διάστημα 2014-2020. Τα τελικά ποσά βεβαίως δεν έχουν ακόμα οριστεί αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ανέλθουν περίπου σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό. Εάν ε, πρόκειται για 3 εκατομμύρια ποσά και πάλι θα χρειαζόμαστε πολύ αυστηρού κανόνε όσον αφορά την χρήση αυτών των κονδυλίων. Αλλά τώρα πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ μεγαλύτερο ποσό Γι' αυτό είναι πολύ δικαιολογημένο όταν πραγματικά κινούμεθα πολύ προσεκτικά, εξετάζουμε τις λεπτομέρειες και ε, αυτή τη φορά προσπαθούμε να είμαστε κάπως κριτικοί αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει ως εξή. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι δοκιμασμένη η λύση να αντιμετωπίσουμε από κοινού την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξη πέθρου. Και νομίζω ότι, ότι εδώ ακριβώς οφείλεται το γεγονός ότι ε, στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής ε, ποτέ δεν έχει τεθεί το ζήτημα η ανάγκη διαχωρισμού αυτών των δύο τομέων. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή αντιμετώπιση αυτών των δύο τομέων είναι χρήσιμη και πάντοτε βεβαίως σε συνάρτηση με την πολιτική συνοχή, όπως είπε και ο κύριος Κρετά. Ε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο συζητούμε συχνά. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περισσότερες περιπτώσεις ε, στο πλαίσιο της νομοθετικής τους εργασίας έχουν σαν σκοπό την απλούστευση των διαφόρων διατάξεων. Βεβαίως ε, θα ήθελα να πω ότι η απλούστευση δεν μπορεί να αποτελεί σκοπό, αυτό το κοπό, αλλά στους περισσότερους τομείς στοχεύουμε παρόλα αυτά σε μια απλούστευση. Οι νομοθετικές προτάσεις παρόλα αυτά είναι πολύ απομακρυσμένες από αυτό το στόχο της απλούστευσης. Πολύ συχνά οι νομοθετικές προτάσεις είναι δυσνόητες, πολύπλοκες, μη εφαρμόσιμες. Αλλά όσον αφορά την εφαρμογή, αυτές οι νέες ε, νομικές διατάξεις πολύ συχνά συνεπάγονται ένα επιπρόσθετο κόστος για τα εθνικά όργανα που επομίζονται με την εφαρμογή τους. Και ε, αφού ε, είδα τι προτάσει για τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργικής πολιτική, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κρετέν όσον αφορά την ανάπτυξη υπαίθρου. Οι διατυπώσει όλες στοχεύουν σε μία πλούστευση. Αλλά ε, στο επίπεδο τη εφαρμογή τελικά θα κάνουν τα πράγματα δυστυχώ πιο πολύπλοκα. Νομίζω λοιπόν ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να έχουμε άκρατο ίνο Δηλαδή να μην μιλούμε συνεχώς για πλούστευση και να κάνουμε στην πράξη το εντελώ αντίθετο. Γιατί μιλάμε μεν για μια πλούστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα ε, δημιουργούμε ένα όλο και πιο πολύπλοκο οικοδόμημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την εξέταση, την παρακολούθηση και σε αυτό αναφέρθηκε η κυρία Ιβάνοβα Νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πιστεύω ότι όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει την αξιοπιστία των εθνικών οργάνων πριν ε, ξεκινήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και εκτός αυτού θα πρέπει να επεξεργαστούμε ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο να είναι γενικά αξιόπιστο. Και τέλος, ε, θεωρώ ότι ένα σημαντικό πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι ότι όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, η στοχοδεσία που έχει διατυπώσει η Επιτροπή ε, αποκλίνει σε πολλές, ε, σε πολλές κατευθύνσεις. Και έχω την άποψη ότι η επίτευξη των στόχων θα πρέπει να τεθεί στο προσκήνιο στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν οι στόχοι θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι πολύ ξεκάθαρα. Αλλά εδώ βλέπω μία αντίθεση. Από τη μία λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μία ξεκάθαρη στοχοθεσία, αλλά από την άλλη έχουμε την πράξη. Γιατί σε ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο όλο δουλειστάνουμε σε συμβασμούς και οι στόχοι ενίοτε είναι αόριστοι. Γι' αυτό ε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ε, διτής διπλής ε, χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν οι στόχοι να είναι εκπεφρασμένοι πιο ξεκάθαρα και πιο εστιασμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρατάν για το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και περιμένω με ανυπομονησία τις πρώτες διαβουλεύσεις σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ήταν μια σειρά από ερωτήματα, αλλά λόγω του μεγάλου καταλόγου των ομιλητών θα σας ε, πρότεινα να δεχτούμε μόνο άλλη μια παρέμβαση, μετά να ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν το είχα καταλάβει ότι θα πάρω το λόγο τόσο γρήγορα. Δεν το φαντάστηκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρετέν. Τον ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κρετέν για την έκθεση αυτή. Όχι μόνο διότι είναι σημαντικότατη, και επειδή ακούσαμε τόσο καλά και κριτικά σχόλια πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί αυτή είναι και η δουλειά του άλλωστε, επίσης όμως διότι τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο βλέπουν το ελεγκτικό συνέδριο σαν κατά ένα καθρέφτη και να αντικαθρεφτιζόμαστε και να βλέπουμε τι κάνουμε. Άκουγα προσεκτικότατα την παρουσίαση του κύριου Κρετέ. Και όλοι παρατηρήσαμε ότι κρύβεται ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και κανείς δεν μιλάει για αυτόν. Γιατί μιλάμε πάντα για τους πόρους και όχι για τους στόχους, για τα αποτελέσματα. Και έχω μια ερώτηση, απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Ελεκτικό Συνέδριο και προς το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη δεν είναι αλήθεια ότι δεν ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα. Ενδιαφέρονται μόνο για τα μέσα, για το σκοπό. Σε κάθε κεφάλαιο σε κάθε πρωτεύουσα, συγγνώμη, από τα 27 κράτη-μέλη, μόνο ένα πράγμα έκαναν. Παίρναν τους υπολογιστές στον ίδιο την πρόταση και έβλεπαν πόσα χρήματα θα τους μείνουν. Ε, το ξέρω, το έγινε στη χώρα μου. Ο Υπουργός Ολλανδός είπε, κοιτάξτε, χάνουμε πολλά, το μόνο που θέλω είναι να μην χάσουμε όσα χάνουμε εδώ πέρα. Ο στόχος που κρύβεται πίσω από την όλη διαδικασία ε, ο τελικό στόχο δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό ο ελέφαντα που στο μισθοδωμάτιο και κανεί δεν τον βλέπει. Δεν ενδιαφέρομαι για τη γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθο. Α είμαστε ειλικρινεί. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συμφωνήσουν με το στόχο της αγροτικής πολιτικής και να μην ασχολούνται μόνο με τους πόρους που ε, χρειάζονται για να πετύχουν το στόχο. Ευχαριστούμε πολύ και θα πρότεινα να, δαθούν, να γίνει ένας γύρος απαντήσεων συγγνώμη, για τις, τις ερωτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις από πλευρά της ηγήτριας της κυρίας Ιβανιώβα όσον αφορά τους φορείς πιστοποίησης και κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μοντέλο όπως το Ταμείο Συνοχής. Πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Χρησιμοποιούμε το ίδιο μοντέλο. Uh, uh, Χρησιμοποιούμε τον ίδιο δημοσιονομικό κανονισμό. που χρησιμοποίησαμε στη Γεωργία είναι το μοντέλο το οποίο τώρα προτείνεται για όλους τους πόρους για την κοινή διαχείριση. Ίσως έχουμε ένα πρόβλημα συνεννόησης εδώ. Ίσως υπάρχει παρεξήγηση αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την κυρία Ιβανούβα και έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο μέλλον και με τον κύριο Κρέτα για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις κυρώσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση, η πολλαπλή συμμόρφωση δεν σχετίζεται με μια πληρωμή που χορηγείται, είναι μια υποχρέωση. Ε, πρέπει να συμμορφωθούν δεόντως οι γεωργοί. Εάν δεν συμμορφωθούν δεόντως επιβάλλεται μια κύρωση. Είναι μια τιμωρία. Μια ποινή. Ένα ποσό που αφαιρείται από οποιαδήποτε πληρωμή που θα λάμβανε κανονικά ο Γιώργος. σύμφωνα με τον ε, κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση αν κατάλαβα την ερώτησή σας το ότι εξαιρούμε μικρούς γεωργού από πολλαπλή συμμόρφωση είναι πολύ οι γεωργοί οι μικροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πρόβλημα για την επίτευξη των στόχων. Θα ήθελα να πω ότι οι μικροί γεωργοί παρόλο που είναι πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι το ποσοστό των γεών που καλλιεργούν είναι μόλις το 3% του συνολικού. Άρα είναι σχετικά μικρό ποσοστό. Γι' αυτό δεν υπονομεύονται οι βασικοί στόχοι των πολιτικών μας. Το ερώτημα του κύριου Ντόιτς αναφέρθηκε στον περίπλοκο χαρακτήρα των προτάσεών μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το εξής. Έχοντας διαφορετικούς στόχους πολιτικών. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα των γεωργών. Θέλουμε να έχουμε καλύτερε συνθήκες για το περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη εδαφική ισορροπία. Και τώρα αυτή είναι απλώ η μεγάλη στόχη αυτή που ανέφερα. Και τα μέσα που διαθέτουμε θέλουμε να είναι τα απλούστερα δυνατά. Αλλά είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε και περαιτέρω απλούστευση. Και θέλουμε να μειώσουμε και το διοικητικό άχθος. Σχετικά με αυτό τώρα. Το 15% αύξηση των διοικητικών δαπανών που ετέθη και συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση αντικτύπου είναι το Ισραίον κόστος για τους γεωργούς και το κόστος που θεωρήσαμε είναι αύξηση του κόστους στη εθνική δίκηση. Το κόστος εισρωών για τους γεωργούς είναι ο χρόνος που πρέπει να σπαταλήσουν για να γεμίσουν τα, τις αιτήσει, δεν είναι πραγματικό κόστος. Και το διοικητικό είναι άλλο θέμα, τούτων λεχθέντων. Ε, έχουμε καταβάλει έκτοτε προσπάθειες για να μειωθεί το διοικητικό αυτό άκθος. Να δώσω ένα παράδειγμα για τους ενεργούς γεωργούς. Επεξεργαζόμαστε πολύ απλουστευμένη προσέγγιση και για τους ελέγχους θέλουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους ελέγχους και για ανάπτυξη της υπαίθρου και για τον πρώτο πυλώνα στον τομέα του πρασινίσματος τη γεωργίας για να μειώσουμε το κόστο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάν Μούλτερ είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επί δύο εκ των τεσσάρων στοιχείων που ανέφερε το ελεγκτικό συνέδριο. Πρώτον, τα κριτήρια για τις πληρωμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι κατάλαβα υπερηφανεύεται κάπως διότι το 2020 οι πληρωμές αναεκτάριο θα είναι πλέον πολύ πιο σώτιμες και ομοιόμορφες στα κράτη-μέλη από ό,τι είναι σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό είναι το σωστό κριτήριο. Προσωπικά πιστεύω ότι η στήριξη του εισοδήματο αναεκτάριο είναι πληρωμή για υπηρεσίες που χορηγούνται στην κοινωνία. Πράσινα, μέτρα πρασινίσματος κλπ. Υποθέτω ότι σε μια περιοχή της Ευρώπης όπου η τιμή ανεκτάριο είναι 50.000 ευρώ, η στήριξη μπορεί, πρέπει να είναι πιο υψηλή από μια άλλη περιοχή όπου η τιμή ανεκτάριο είναι 5.000 ευρώ. Διότι εξορισμού, αν είναι ακριβή η γη, κοστίζει περισσότερο να εφαρμόσει κανείς περιβαλλοντικά μέτρα από εκεί που είναι πιο φθηνή η γη. Σε ποιο βαθμό το παίρνει υπόψη της αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αυστηρά κριτήρια για να κρίνει και να πει αυτή είναι μία πληρωμή που δικαιολογείται σε αυτές τις περιοχές. Και αν το κάνει αυτό, βάσει ποιων κριτηρίων κρίνει. Δεύτερον, οι φορείς πιστοποίησης έχουν πολύ λιγότερο σημαντικό ρόλο, μειώνεται η σημασία, καλώς, όμως η έγκριση των φορέων πιστοποίησης ε, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστεύεται τους φορείς πιστοποίηση, θα πρέπει να τους εγκρίνει επίσης. Και γιατί δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που έχω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος, κύριος. Uh, Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πριν θέσω το ερώτημα να πω κάτι για να προετοιμάσω το έδαφος για την ερώτηση. Είμαι νέος εδώ, αλλά κάθε πρωί προσπαθώ να θυμηθώ κάτι. Γιατί είμαστε εδώ. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με αυτό που θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μιλάμε για 300 δις ευρώ, και το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ πολιτών και Ευρώπης και πώς βλέπουν το όλο πράγμα, διότι η Γεωργία είναι κατά πολύ το μεγαλύτερο κομμάτι. Και τι περιμένουν από μας παραγωγικότητα περιμένουν. Όλη η μέρα, χτες και σήμερα, ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας και σας προειδοποιώ για κάτι, εκ των προτέρων προειδοποίηση. Απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πάνε στη, στο Συμβούλιο Γεωργία και πούν ο, ή στην Επιτροπή Γεωργία και πούν ότι εν είδη απαντήσω προ τον κύριο Κρετά και το έργο του και πούν ότι προσπαθούν να καθορίσουν ποιος είναι ο ενεργός γεωργός. Και όταν βρουν περί τίνος πρόκειται, τότε θα επεξεργαστούν τους ελέγχους βάση τουρισμού να σας πω ότι η Επιτροπή Γεωργίας δεν θα το ανέχθει αυτό, δεν το δεχτεί αυτό, δεν το καταπιεί. Διότι είναι ξεκάθαρο το θέμα για αυτούς. Αυτό δεν θα το δεχτούν στις μεταρρύθμιση. Λοιπόν, να πω κάτι με κριτικό πνεύμα. Αφορά το πώς εξετάζουμε το θέμα, πώς το προσεγγίζουμε. Και λέω, Δεν πρέπει να μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες και στα θεωρητικά επιχειρήματα. Τι είναι ενεργός γεωργός. Δεν υπάρχει ορισμός και δεν θα υπάρξει ποτέ συμβιβασμός. Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκάιερ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ναι, θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής και θα συνεχίσω εδώ βεβαίως ε, πρόκειται για μια πολιτική σύγκρουση αλλά θα πρέπει για μια φορά να το ρισκάρουμε εν ανάγκη δηλαδή υπολογίζεται στην ε, Επιτροπή ε, ότι η Επιτροπή Γεωργίας δεν έχει πολύ πλατιά υποστήριξη. Εγώ, σοσιαλδημοκράτης, χαίρομαι που οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Γεωργίας έχουν ε, προχωρήσει τόσο πολύ που δέχονται να περιοριστούν οι ενισχύσεις τους λεγόμενους ενεργούς γεωργούς. Δηλαδή οι ενισχύσεις εφόσον ε, πρόκειται το τεράστιο μπλοκ της γεωργίας ε, δεν μπορούν να είναι λιγότερες αλλά τουλάχιστον να είναι στοχευμένες, επικεντρωμένες. Γιατί εμείς εδώ ε, προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε μια γεωργική πολιτική η οποία φτάνει στον ε, καλλιεργητή. Ένα από τα πιο, μια από τις πιο αποκτές ε, στιγμές στον πολιτικό μου βίο ήταν όταν έλαβα μέρος σε μια διάσκεψη για τη Γεωργία και τελικά διαπιστώθηκε αυτό το οποίο είπε η προηγούμενη ομιλήτρια ε, δηλαδή ποιο είναι τελικά το μέλλον της γεωργίας και ε, όλες οι ανησυχίες των 17 ε, υπουργών γεωργίας ήταν πώς μπορούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα ή πόσα χρήματα θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανείς δεν έφεσε το ερώτημα για ποιο σκοπό. Και όταν κάποιος είπε ότι ένας μηχανισμός όπου δεν διενεργείται κανένας έλεγχος ε, γιατί μπορεί να πρόκειται για ένα γήπεδο γκολφ τελικά ή ένα χέρσο κομμάτι το οποίο απλώς στηρεί τις περιβαλλοντικές ε, περιγραφές. Ε, τελικά το αντεπιχείρημα ήταν ότι με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται η θέση της Γερμανίας εάν ε, γύρουμε τέτοια ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ενισχύει την κοινή γεωργική πολιτική, ούτε μπορεί να κερδίσει την ε, συγκατάθεση των Ευρωπαίων πολιτών για το πού πάνε τα... για σκοπούς με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα χρήματά τους. Ε, δεν είναι δυνατόν να καταλήγουν ε, τα χρήματα αυτά οπουδήποτε, αρκεί να τρέχει κάνουλα. Γι' αυτό υποστηρίζω τις προσπάθειες της Κομισιόν τελικά τα κονδύλια αυτά να φτάνουν στους ε, γεωργούς και όσο πιο στοχευμένα χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά, τόσο πιο εξασφαλισμένα θα πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλη μια παρέμβαση και θα κλείσουμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφος κύριος Λιμπεράτσκι θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική γεωργίας είναι ο τομέας όπου ποσοστιαία έχουμε τα περισσότερα κονδύλια στον προπολογισμό. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας, γιατί το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο στηρίζουμε τους παραγωγούς ή τελικά τους καταναλωτές. Και δεύτερον, το θέμα είναι κατά πόσο στην ε, ε, παγκόσμια αγορά για τα γεωργικά προϊόντα ε, μπορούμε να έχουμε μια ελευθερία ή θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποιους κανόνες που επιβάλλονται έξωθεν. Και η απάντηση είναι ότι συγκεντρωνόμαστε κυρίως στον πολίτη για το πρώτο ερώτημα και δεύτερον πρέπει να προσανατολιστούμε προς τα πράγματα τα οποία χρειάζονται οι εταίροι μας. Τρίτον, δεν θα πρέπει να χάσουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα μεταποιούμε. Γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις εισαγωγές τροφίμων ή και t-shirts. Αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η εξάρτηση από τις εισαγωγές όσον αφορά τα τρόφιμα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είναι μια νέα χώρα, ένα νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε γνωρίσαμε καλύτερες ε, μέρες. Και αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα, γιατί οι άμεσες ε, γιατί η αναδιάρθρωση τελικά υποστηρίζει ορισμένες ομάδες πολιτών και αυτό οδηγεί σε μια συγκέντρωση της ε, παραγωγής καθώς και της ιδιοκτησίας γης. Είναι γεγονός ότι η συνέχιση της ε, παρούσας κατάστασης θα απολυθώσει τις ε, υφιστάμενες δομές. ναι, λένε ότι βρούνται θέσει απασχόληση, αλλά από την άλλη, αν δεν αυξήσουμε τι άμεσε ενισχύσει, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να φύγουν πολύ από τη χώρα, να εγκαταλείψουν τη χώρα, την ύπεθρο χώρα. Και ήδη έχουμε 30% ανεργία. Και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση αυτών των αριθμών. Το ερώτημα είναι λοιπόν κατά πόσο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο είδου κίνητρο σε μια περίοδο κρίσης όπου η έξοδος από την κρίση ε, δεν είναι ορατή. Θα πρέπει να επιδεινώσουμε ακόμα τα ποσοστά της ανεργίας ή θα πρέπει να κοιτάξουμε να αυξήσουμε τις άμεσες ενισχύσεις. Παρόλο που ο κύριος ε, Μούλτερ τάχθηκε κατά αυτής της δυνατότητας. Και βεβαίως υπάρχει το κριτήριο των ε, τιμών των διαφόρων γεωργικών ε, εκτάσεων. Ε, Βεβαίω αυτό συνδέεται και με την παραγωγικότητα. Ο κύριο Γκάιερ θα το ερώτημα το πώ μπορούμε αυτό να το διανύμουμε, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά γεωργίας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και πάλι ήταν μια, ένα ολόκληρο πακέτο ερωτήσεων. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πατσέκο να πάρει θέση εξ ονόματος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτον, η ερωτήση του κυρίου Μόλιντερ. Λοιπόν, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ισχύον σύστημα βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Βασίζεται στο τι Στι, στις παρελθούσες δηλαδή συγκομιδές παραγωγές του Γεωργού. Και οι πιο παραγωγικές χώρες είχαν υψηλότερους συντελεστές. Είναι δικαιότερο αυτό το σύστημα ή αυτό προς το οποίο κατευθυνόμαστε. Όχι είναι η απάντηση κατά τη γνώμη μας. Θέλουμε να εγκαταλείψουμε τα ιστορικά μοντέλα μου θέσατε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ποια ακριβώς είναι τα εφαρμοστέα κριτήρια για τη σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε ακριβώς κριτήρια, έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Και νομίζω είναι, ότι είναι ένα χρήσιμο στοιχείο στα πλαίσια της συζήτησης για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και σε κάθε περίπτωση... Μας επιτρέπει αυτό το σύστημα να υπάρξει σύγκληση των ενισχύσεων προς τα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν είναι άλμα, αλλά είναι ένα μικρό βήμα σε κάθε περίπτωση προς τη σωστή κατεύθυνση και εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση περί ανακατανομής των κονδυλίων. Για τους ε, φορείς επιστοποίησης, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ανεξάρτητους φορείς που ακολουθούν δικά τους ανεξάρτητα ελεγκτικά πρότυπα. Αυτά τώρα ε, στο, στα πλαίσια της ε, μικτής ε, συνδιαχείρισης, της κοινή διαχείρισης, της συνδιαχείρισης ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα ήθελα για 30 δευτερόλεπτα να μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ στο θέμα του ενεργού γεωργού. Άκουσα εδώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η έννοια, διότι πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς γεωργούς. Αυτό είναι σωστό, αλλά καταλαβαίνω και τον σκεπτικισμό που υπάρχει σε σχέση αν θα το καταφέρουμε το στόχο μας χρησιμοποιώντας τον ορισμό που προβλέπεται. Με την ΚΟΜΑΓΡΕ συνεργαζόμαστε και ευελπιστούμε να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό, ώστε να καταλήξουμε, πώς να το εξηγήσω, σε ένα διπλό σύστημα. Πρώτον, δεν χορηγείται ενίσχυση σε έκταση που δεν είναι έτοιμη για γεωργική χρήση ή που δεν χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. Δεύτερο κριτήριο αρνητικό, δεν θα δώσουμε ενισχύσεις για γήπεδα του γκολφ παραδείγματος χάρη για οποιασδήποτε αθλητικές δραστηριότητες σε ρολιμένες κτλ. Ε, ένας αρνητικός κατάλογος δηλαδή. Μόνο στην περίπτωση όπου θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει ε, εσφαλμένη καταβολή ενίσχυσης, θα πρέπει εκείνος να αποδείξει ότι ε, η εκμετάλλευσή του έχει γεωργικό χαρακτήρα και ότι, δεν, ε, και ότι το 95% είναι για γεωργική χρήση. Το βάρος της απόδειξης βαραίνει τη δεύτερη κατηγορία, τον αρνητικό κατάλογο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι η κόμμα Αγκρή, συνάδελφοι από την κόμμα Αγκρή και εγώ πιστεύω ότι έτσι θα ε, καταφέρουμε να επιτύχουμε καλύτερα το στόχο μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πατσέκο για τις απαντήσεις σας. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, ε, ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. Θα διευκρινίσω, δεν ήμουν ξεκάθαρος μάλλον, να σας πω τι εννοούσα. Εάν αυτό είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που θα δώσετε στην Επιτροπή μας για να αποδείξετε ότι υπάρχει αυστηρότερη διαχείριση ε, των πόρων ε, δεν ε, έχει πολύ ψαχνό. Καταλαβαίνετε, πείτε μας, δώστε μας κάτι καλύτερο. Αυτό εννοούσα πριν. Μάλιστα. Η διευκρινιστική ήταν αυτή η παρατήρηση, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εάν το επιθυμεί ο πρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο κύριος Κρετά μπορεί να ξαναπάρει το λόγο για να κλείσει και η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Αφήστε που ελάχιστες ερωτήσεις απευθύναν οι συνάδελφοι στο ελεγκτικό συνέδριο για τις διευκρινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τον όλο προβληματισμό και διάλογο για τον ε, ενεργό γεωργό έχει, έχουν ιδιαίτερη σημασία, ε, το αναγνωρίζω, αλλά αντίθετα δεν ικανοποιήθηκα από τις διευκρινήσεις κάποιων επιμένους διατάξεων που είναι απαραίτητες, συγκεκριμένα για τον ρόλο των οργανισμών πιστοποίησης την ε, ε, σημασία και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 97, σας τα έλεγα και προηγουμένως, και το θέμα των ε, καταποκοπήν διορθώσεων. Ξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για αυτές τις κατακοπήν ε, διορθώσεις ε, ανάμεσα στον γεωργικό κανονισμό και τον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Α, μόνο, όπως σας έλεγα και το πρωί, στις 4.30 πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην Επιτροπή Γεωργίας και άρα θα πρέπει να αποχωρήσω. Ευχαριστούμε και καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. νομίζω ότι είναι μια καλή χρονική στιγμή, γιατί όπως ανέφερε ο κύριος Κρετάν στο τέλος, η συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική τώρα έχει πάρει μια σωστή όφηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο υπαριθμών 3, ή μάλλον το ε, Ηρακλής 3. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ιβάνοβα. Και εδώ υπάρχει ένα κείμενο εργασίας, ένα έγγραφο εργασίας του ελεγκτικού συνεδρίου Äh, äh, äh, κύριο Τσβίκελ είναι αρμόδιος και θα ήθελα να παρακαλέσω καταρχήν την εισηγήτρια να μας κάνει μια παρουσίαση και στη συνέχεια θα ήθελα να χαιρετήσω από την Όλαφ τον κύριο Γκάους και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τον κύριο Τσβίκελ πριν ακούσουμε από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού τον κύριο Ταβέρν. Παρακαλώ, κυρία Ιβάνοβα, εφόσον το επιθυμείτε. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα παρουσιάσω αυτό το πρώτο έγγραφο εργασίας, το οποίο αποτελεί μόνο μια εισαγωγή στο όλο θέμα. Τι, ο Ηρακλής για τι πράγμα είναι. Δημιουργήθηκε σαν ειδικό πρόγραμμα δράσης κοινοτικό για την πρόθεση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Το 2004 δημιουργήθηκε. Είχαμε το Ηρακλής 1 και 2 και τώρα αυξήθηκε το πεδίο εφαρμογή του Ηρακλής 2 για να χρηματοδοτήσει και δραστηριότητες που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης και λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Στο Ηρακλής 3 που θα συζητήσουμε σήμερα συνεχίζουμε την επιδίωξη των λόγων στόχων το παρόν πρόγραμμα Ερακλής 2 λύγει το Δεκέμβριο 2013. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε το παρόν πλαίσιο και πόσο αποτελεσματικό ήταν το πρόγραμμα και να εξασφαλίσουμε τη συνέχισή του. Το νομικό και οικονομικό πλαίσιο που υπάρχει τώρα αφήνει διάφορα ερωτηματικά, διάφορε εκκρεμότητε θα πρέπει να καλυφθούν στα πλαίσια τη εγκρίσεω των νομοθετικών πράξεων. Είναι το πρώτο από τα δύο έγγραφα που θα εστιάζονται επί τριών σημαντικών θεμάτων που θεώρησε ότι σε αυτή τη φάση πρώτα απ' όλα είναι πρώτα απ' όλα η προσημείωση και συντονισμός, δεύτερον αξιολόγηση των προγραμμάτων και μετά ε, διαχείριση των προγραμμάτων και αποτίμηση, αξιολόγηση. Να πω σαφώ ότι το Κοινοβούλιο και ιδίως αυτή η Επιτροπή πάντα υποστήριζαν ένθερμα την καταπολέμηση των λαθρεμπορίου σιγαρέτων και των παραποιημένων προϊόντων αδιαμφισβήτητο αυτό. Το ερώτημα που θέτω σήμερα είναι πόσο αποτελεσματικές είναι οι δαπάνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως για αυτούς τους σκοπούς και αν μπορούμε να είμαστε πιο συντονισμένοι, να συντονιστούν καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να καταλήξουμε και σε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων και του λαθρεμπορίου. Χαίρομαι που έχουμε τον Γκιότ Σφίκελ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί μα, Έχουμε την Όλαφ, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μοιραστούν μαζί μας ε, τις δικές τους απόψεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρώτο θέμα όσον αφορά την προσημείωση, earmarking. Το πρόγραμμα Ηρακλής 3 θα εξακολουθεί να υποστηρίζει δαπάνες που σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Αυτός ο στόχος θα πάρει το σημαντικότερο ποσό από 98,6 εκατομμύρια ευρώ του Ηρακλής 2 θα πάει στα 110 εκατομμύρια ευρώ στο Ηρακλής 3. Φαίνεται ότι διάφορα θεσμικά όργανα έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αρχή της καθολικότητας και εγώ προβληματίζομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πράγματι διατηρείται η αρχή της καθολικότητας όταν συνεχίσουμε με το Ηρακλής η Όλαφ φαίνεται ότι πιστεύει ότι η αρχή της καθολικότητας εφαρμόζεται και αναφέρει ότι το Ηρακλή 3 με του πόρους του μπορεί να αφιερωθεί σε δραστηριότητε που αφορούν την καταπολέμηση λαθρεμπορίου σιγαρέτων και παραποίησης προϊόντων. Πιστεύω όμω ότι χρειαζόμαστε ανοιχτή πραγματική συζήτηση με συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να ακούσω και τι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού καθώς και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το δεύτερο θέμα αφορά τη βιωσιμότητα της χρηματοδοτήσεως και την πρωτοβουλία κατά του λαθρεμπορίου, πρωτοβουλίες μάλλον, και συντονισμός που πρέπει να υπάρχει μεταξύ δραστηριοτήτων Όλαφ και δραστηριοτήτων κρατών μελών. Σε αυτή τη φάση δεν είχαμε αρκετέ πληροφορίες όσον αφορά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ηρακλής και του Ηρακλής 2 δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πώς ακριβώς δαπανήθηκαν τα ποσά, ποιο συντονισμός υπήρξε ε, με τις εθνικές πρωτοβουλίες, ούτω ώστε όλες αυτές οι προσπάθειες που καταβάλλονται να δικαιολογούνται πραγματικά και να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων. Να μην επαναλαμβάνεται κάτι που κάνει τα κράτη-μέλη και να ξοδεύει λεφτά και η παράλληλα το θέμα της αξιολογήσεως του προγράμματος. Πάνω σε αυτό είχαμε γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου το 2006 και ειδικέ εκθέσεις. Βασικά πορίσματα ποια είναι ότι όπως και σε άλλους τομείς μας, λείπει, μας λείπουν σαφείς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων αυτό αναφέρεται και σε δύο έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξολόγηση αντικτύπου και η ενδιάμεση αναθεώρηση το ανέφεραν. Έθεσαν και το θέμα των στόχων του Ηρακλής 2, την ποιότητα των δικτών που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και τη νέα περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί κάποιου δείκτε, όπω το ποσό των ανακτήσεων, η αύξηση του ποσοστού των κοινών επιχειρήσεων, η αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που αποδέχεται αποδέχονται οι, ποινικές, οι αρχές της ποινικής δίωξης για να εφαρμόσουν τους στόχους του προγράμματος. Οι δείκτες δεν καλύπτουν όμως όλες τις δραστηριότητε για τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν. Όπως κατάρτιση, οι διασκέψεις. Δεν έχουμε δείκτες επιδόσεων για να προσμετρήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Χρειαζόμαστε όχι μόνο ποσοτικά αποτελέσματα και εκροές, αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα. Θέλουμε να μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τέλος, εξίσου σημαντικό, το θέμα της διαχειρίσεως των προγραμμάτων και της αξιολογήσεως. Καλωσορίζω δύο επιτεύγματα. Πρώτον, δημιουργήθηκε ενιαία μονάδα της OLAF, η οποία θα συντονίζει τη διαχείριση όλων των δράσεων που σχετίζονται με κοινοτικά προγράμματα στον τομέα τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη κοινότητα Θα βελτιώσει επίση την ενοποίηση και εναρμόνιση των διαδικασιών των εφαρμοστικών μεταξύ όλων των τομέων χρηματοδοτήσεως και θα δημιουργηθεί και νέα εσωτερική βάση δεδομένων που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Όλαφ Έχω ένα ερώτημα όμως, ένα θέμα που συζητήθηκε στην ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2011 και αφορά το θέμα της εγχειρήσεως των προγραμμάτων και ενδεχόμενο συγκρούσεως συμφερόντων. Να είναι αποδέκτης και διαχειριστής και ελεγκτής όλα αυτά ταυτόχρονα και χρήστης των πόρων. Θα ήθελα να ζητήσω από την Όλαφ να το σχολιάσει. Θα ήθελα να ακούσω επίσης τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να δω πόσο καρποφόρο θα είναι η συζήτησή μας. Περιμένω να ακούσω τα σχόλια της Όλαφ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάνω απ' όλα τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Yeah, thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Ιλιάνα. Πολλά σημεία έθεσες. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Όλαφ. Δεν είμαι σίγουρος αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ο κ. Κάουφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Συγήτρια, κυρία Ευανόβα για τα διευκρινιστικά σας σχόλια. Ευχαριστώ σας και το έγγραφο εργασίας που έχει συνταχθεί. Θα δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για την προσημείωση των ποσών. Όσον αφορά κάποια από τα στοιχεία που θίξατε, πράγματι μπορούμε να σας δώσουμε τις εξής πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα σχετικά με το Ηρακλής 2, το τρέχον πρόγραμμα Ηρακλής, το οποίο φτάνει μέχρι το 2013 στις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Σας έχουμε δώσει την ενδιάμεση ανεξάρτητη αναθεώρηση του Ηρακλής 2, συνετάχθη το 2010 από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Όλαφ και δίνει αρκετά λεπτομερή επισκόπηση των δράσεων που διενεργήθησαν στα πλαίσια του Ηρακλής 2 κατά την περίοδο που εξετάζουμε. Τρία χρόνια αξιολογήσεως με άλλα λόγια. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Πολλά προγράμματα τεχνικής αρρωγής για υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη ε, εφαρμόστηκαν αγοράστηκαν σαρωτές, συμφωνίες με διάφορες αρχές για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου σιγαρέτων, πράγματος χάρη, η ενδιάμεση εξολόγηση συνεπιών, στην οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 η απόφαση για το Ηρακλής 2, δίνει αρκετά σαφή εικόνα των όσων συνέβησαν, των αποτελεσμάτων των δικτών που χρησιμοποιήσει η Όλαφ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τη εφαρμογή του Ηρακλής 2. Άρα είναι πολύ χρήσιμο το έγγραφο για περαιτέρω συζητήσει περί των επιτευθέντων αποτελεσμάτων. Βέβαια, κάναμε μια περίφημη διαβόητη αξιολόγηση συνεπειών ετοιμάζοντας την πρότασή μας, την οποία υποβάλαμε στην νομοθετική αρχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλοι έχετε την αξιολόγηση συνεπειών ΚΟΜ 2011-914, αξιολόγηση αντιχτυπου Εκεί τονίσαμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Επικαιροποιείται η ενδιάμεση αναθεώρηση που εξεπώνησε η μονάδα μας εσωτερικού ελεγχού. Αξιολόγηση συνεπειών λοιπόν και η δήλωση νομοθετικού περιεχομένου και το σχέδιο κανονισμού η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερόταν σε κάποιους δείκτες επιδόσεων αποτελεσμάτων. Θέλουμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες περισσότερο όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο στοιχεία γι' αυτό. Πρώτον, χρειάζεται γενική τελική αξιολόγηση του Ηρακλής 2 πριν το τέλος 2014. Βάσει της τελικής αξιολογήσεως των αποτελεσμάτων του Ηρακλής 2 θα ετοιμάσουμε προτάσεις για πιο συγκεκριμένους δείκτες που θα ευθυγραμμίζονται με τους δείκτες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να είναι πιο περιορισμένη η ερμηνεία. Θέλουμε πιο ποιοτικού δείχτε, όχι τόσο ποσοτικού όσου έχουμε, τώρα, όσους έχουμε τώρα. Μετά, όπως υπόθηκε και αναφέρεται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπαμε ότι θα συζητήσουμε το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το Ηρακλής 3 στο μέλλον στην ομάδα εμπειρογνωμόνων κατά της απάτης στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Κόκολαφ. Εκεί θα συζητήσουν τις προσωπίες και τις εμπειρογνώμες των κρατών μελών, το ετήσιο πρόγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει να προσμετρηθούν αυτά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσουμε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για συζητήσεις για ενδεχόμενους δείκτες επιδόσεων. Τέλος, εξίσου σημαντικό. Όταν εφαρμόζουμε το Ερακλής 2 τώρα, χρησιμοποιούμε ετήσιες αποφάσεις χρηματοδοτήσεων που είναι προϋπόθεση σύμφωνα με τον οικονομικό Κανονισμό. Παρουσιάζουμε πρόγραμμα εργασιών, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε κάποιο βαθμό αναφέρεται σε δείκτες επιδόσεων. Και όλες αυτές οι προσεγγίσεις θα συζητηθούν και στην ομάδα εμπειρογνωμών στην Κοκόλαφ. Μαζί με τα κράτη-μέλη, όπως σας προανέφερα και επαναλαμβάνω και τώρα. Για να συζητήσουμε τους δείκτες επιδόσεων. Και για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις δράσεις που προγραμματίζονται και αυτές που εφαρμόζονται. Αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζω ότι μπορούμε να σας δώσουμε και οι πληροφορίες να δίνουν κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις που ετέθησαν στην παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσφίκελ τώρα από το ελεγκτικό συνέδριο θα κάνει τη δήλωσή του. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, εκπονεί τώρα την γνωμοδότησή του για το ε, Ηρακλής 3 ε, και συζητούμε τα θέματα και με την κυρία Ιβάνοβα. Η κυρία Ιβάνοβα εξάλλου έκανε και πρώτη ανταλλαγή απόψε με την Όλαφ και στο τέλος τη τρέχουσα εβδομάδα έχει προβλεφθεί άλλη σύσκεψη. Τέλο πάντων, θα ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μα σύντομα. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μας, δεν έχει εγκριθεί ακόμη η γνωμοδότηση, οπότε με την ιδιότητα του μέλου του ελεγκτικού συνεδρίου το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να υποδείξω τις γενικές γραμμές που θα ακολουθήσει η γνωμοδότησή μας. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένα πορίσματα, τέλο πάντων. Και συνοπτικά θα έλεγα ότι τα βασικά ζητήματα που εντοπίζουμε στην γνωμοδότησή μας ε, είναι παρεμφερή με αυτά που αναφέρει η συγγήτρια στα έγγραφα εργασίας του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ε, γενικόλογες παρατηρήσεις και κάποια πιο ειδικά σχόλια. Πρώτον, η μεταξέλιξη του Ηρακλής 2. Ε, έχουν δοθεί πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό έχουν ε, ολοκληρωθεί τα προγράμματα του Ηρακλής 2. Θέλουμε λοιπόν από πλευρά τη Όλευση Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία απάντηση. Έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στόχοι του Ηρακλής 2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο 1η Πρώτου 2007 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 και αναρωτιόμαστε το εξής. Προτού ε, αρχίζει το Ηρακλής 3 ε, δεν θα έπρεπε να καταδείξουμε ότι με αυτά τα πρόγραμματα έχουν επιτευχθεί ήδη οι στόχοι του Ηρακλής 2. Δεύτερη γενική παρατήρηση. Αυτό συνδέεται με τα κονδύλια τα εθνικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την καπνοβιομηχανία. Περίπου 40% του προγράμματος Ηρακλής 3 ε, 44 περίπου εκατομμύρια διοχετεύονται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Αυτό απηχεί την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προκύπτει από τη Διεθνή Συμφωνία των Καπνοβιομηχάνων για το θέμα αυτό. Παρόλα αυτά, 90% και πάνω των 9 δις ε, από το 2004 μέχρι το 2008 προέρχεται από τον εθνικό προϋπολογισμό και εφόσον 90% τη συμφωνίας ε, σχετίζεται με τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη, θα επιζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της κατάστασης, ούτως ώστε να αποφύγουμε την επικάλυψη της χρήσης των εθνικών κονδυλίων βάσει της συμφωνίας. Στο σχέδιο γνωμοδότης αναφερόμαστε ε, στην ανάγκη για ε, μεγαλύτερη ενημέρωση σε σχέση με τα κονδύλια που υπάγονται σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό θα πρέπει να μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουμε μια ενιαία και συντονισμένη προσέγγιση για τη χρήση των πόρων και πάνω από το μισό των δύο δις ε, σύντομα θα έχουν δαπανηθεί και ε, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να καταλάβουμε αν έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στόχοι του Ηρακλή 2. Κάτι άλλο σχετικό με το ε, Ηρακλή 3 και τις ε, συμφωνίες ε, με τις καπνοβιομηχανίες έχει σχέση με το ενδεχόμενο κενό χρηματοδότησης. Εκπνέει το 2016 μία από αυτές τις συμφωνίες και άρα θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η πρόθεσή της, να παρατείνει ε, τη συμφωνία ή να ε, ασχοληθεί γενικότερα με το σε εισαγωγικά κενό χρηματοδότηση για τα προγράμματα Ηρακλήστρια. Θα βρει μια εναλλακτική λύση. Τέσσερις ε, ειδικέ παρατηρήσεις. Πρώτον, αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιέφερε μάλλον η αιτιολόγηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη πρόταση περί αυξήσεω του ποσοστού συγχρηματοδότηση από τα 50 ε, στα 80% και σε ορισμένε ε, αιτιολογημένε περιπτώσει μέχρι και 90% θα είναι το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Πιστεύω ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί ισχύουν και για τον προπολογισμό τη Ένωση. Δεν γνωμοδοτούμε εδώ, το τονίζω. Θέλουμε περισσότερα στοιχεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν, διαχείριση της Όλαφ για το πρόγραμμα Ηρακλής 3. Σε μια πρόσφατη έκθεσή μας για την Όλαφ κάναμε το εξή σχόλιο. Η Όλαφ θα έπρεπε να εστιάσει τις δραστηριότητες της στον ερευνητικό της ρόλο και όχι να διαχειρίζει προγράμματα ε, προϋπολογισμού όπως το Ηρακλής 2 ή 3. Περιμένουμε την απάντηση στην Όλαφ και θα επανέλθουμε σε αυτό στην επικείμενη γνωμοδότησή μας. Τέταρτον. Δείκτες αποδόσεως. Όπως ε, το αντιλαμβανόμαστε τώρα, δεν είναι πολυμετρήσιμοι αυτοί οι δείκτες. Δεν προσδιορίζονται επακριβώς. Και αυτό θέλουμε να το συζητήσουμε με την Όλεφ. Τέλος. Όντως προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία ε, για προγράμματα για ενισχύσεις κάτω από 50.000 ευρώ, αλλά όλα αυτά είναι συνάρτηση του κανονισμού περί εφαρμοστικών διατάξεων που τώρα διαπραγματεύεται. Η Επιτροπή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αυτές είναι οι αρχές μας σκέψεις ε, και περιμένουμε την συζήτηση που θα γίνει και τις επαφές ε, που θα κάνουμε, ούτως ώστε τέλη Ιουνίου περίπου να ολοκληρώσουμε την ε, γνωμοδότησή μας και φυσικά θα επανέλθουμε εδώ στην Επιτροπή σας, ε, αν το επιθυμείτε φυσικά, για να σας παρουσιάσουμε στο ακεραιό της τη γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε κυρία Τσίκλε. Και ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ταβέν από την Επιτροπή για να τοποθετεί πριν μπούμε στην ε, συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα εισοδήματα που έχουν αποδοθεί υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα θέμα αρχής ε, και επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού να γίνει απολύτως σεβαστή. Σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, στα, στον τελευταίο τριμερή διάλογο καταλήξαμε ε, σε μερική συμφωνία περί του άρθρου 18 του, σχεδίου, του νέου σχεδίου δημοσιονομικού κανονισμού. Όμως, ε, ε, θέλει να, εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει ένα μέρος των εσόδων η Επιτροπή από τις καπνοβιομηχανίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, διότι αν ανοίξουμε το παράθυρο για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος υπεράσπιση οικονομικών συμφερόντων, αναπόφευκτα θα προσπαθήσουν και άλλοι να υποφεληθούν από αυτήν την πηγή εισοδήματος για άλλα προγράμματα, όπως για τις κοινωνικές παροχές ή προγράμματα στον τομέα της ε, υγείας ε, και άρα θα πρέπει να μοιράσετε την πίτα σε περισσότερους. Θα βρεθείτε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και θα έχετε ανοίξει και το κουτί της Πανδώρας. Υπάρχει ένα άλλο τώρα ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα επιχείρημα. Αυτά τα ποσά δεν μπορούν να απορροφηθούν από τα προγράμματα γιατί παρά είναι υψηλά. Τι γίνεται λοιπόν. Το earmarking, εν τη αυτή περίπτωση, θα λειτουργήσει αντικά. Δηλαδή θα ε, δεσμεύουμε υπερβολικά πολλά ε, κονδύλια για ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Γι' αυτό και έκανε δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανέλαβε τη δέσμευση να εισηγηθεί στι αρχέ ε, αρμόδιες για τον προπολογισμό κάθε έτος μέχρι το 2020 ένα ποσό θα προτείνει ένα προϋπολογισμό δηλαδή, για να αποφασίσουν οι αρχές που είναι για τον προϋπολογισμό. Αλλά ε, θα συζητάμε τις πιστώσεις πληρωμών και όχι τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Ε, επί τη βάση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποφασίζει λοιπόν η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και έτσι θα ε, γίνει σεβαστή η αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού. Αυτή η θέση θα εγκριθεί στη διυπηρεσιακή σύσκεψη την Πέμπτη την Παρασκευή, αλλά πάντως οι αρχές μου με διαβεβαίωσαν ότι θα υιοθετηθεί αυτή η θέση όπως ε, σας την περιέγραψα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Κύριε Μπαλτσίτη, εσείς θέλατε να πάρετε το λόγο. Θα ήθελα να πάρω θέση για αυτό το θέμα, γιατί στη Λιθουανία εδώ και 15 χρόνια δράει Φίλιπ Μόρις και υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη χώρα μας. Έχουμε σύνορα με την Ρωσική Ομοσπονδία, τη Λευκορωσία και το Ηρακλής 2 και 3 δεν θα διακριθούν, δεν διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενό τους. Ίσως θα αλλάξουν οι βασικές αρχές του ελέγχου, αλλά έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ και σχετίζονται με ένα προϊόν το οποίο εξασφαλίζει πάρα πολλά έσοδα στους προπολογισμούς. Τελευταία είχαμε μια επίσημη πληροφορία ότι μέχρι ε, ότι πολλούνται έως και 43% παράνομα τσιγάρα, τα οποία περνάνε παράνομα τα σύνορα και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα Ηρακλής και ε, ε εφόσον συζητούμε για τις βασικές αρχές του προγράμματος θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Όλαφ και τις άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν ε, συλλέξει μια πλούσια εμπειρία στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με εκείνες τις χώρες όπου οι τιμές ε, των σιγαρέτων είναι κατά πολύ χαμηλότερες λόγω του φορολογικού συστήματος και λόγω άλλων παραγόντων. Γι' αυτό το λόγο ε, εγώ τάσομαι υπέρ μια συνέχισης του προγράμματος και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότερα κονδύλια για τον ε, απαραίτητο εξοπλισμό, για τη δημιουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων ούτως ώστε να μπορούν να ανοιχνεύονται τα παράνομα τσιγάρα μέσω δορυφορικών προγραμμάτων ή συστημάτων πλοήγησης. Ε, εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό ασφαλώς θα εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα τόσο στις χώρες μέλη. Ε, ε, στις χώρες μέλη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαλτσίτο, κύριος Γκάιρα. Ähm, wir haben als fraktion überhaupt keine Ως ε, σοσιαλιστική ομάδα δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τα θέματα τα οποία έθεσε η κυρία Ιβάνοβα, αλλά θα ήθελα να εμπλουτίσω τη συζήτηση φέρνοντας ένα άλλο θέμα. Εάν δω τις νομικές πτυχές, οι χώρες μέλη είναι βάσει της συνθήκης αρμόδιες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την παρεμπόδιση του λεφερμπορίου τσιγάρων. Και μόνο η Τσεχία δεν έχει κυρώσει αυτή τη συμφωνία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η νομική κατάσταση. Τώρα βεβαίως ε, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου το Συμβούλιο ταυτόχρονα ε, είναι το ίδιο θεσμικό όργανο και λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για προστασία των εξωτερικών συνόρων που ε, μας υποχρεώνει η συνθήκη ε, θα θέλαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα από τον κοινό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να είμαστε καλύτερα σε θέση αυτό να εκπληρώσουμε το έργο το οποίο μας αναθέτει η συνθήκη. Άρα λοιπόν έχουμε μία μετατόπιση των κονδυλίων από τους εθνικούς προπολογισμούς, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα έχουμε την κατάσταση το Συμβούλιο άλλων χωρών μελών, αλλά το ίδιο θεσμικό όργανο παρόλα αυτά, να πει ότι ε, θέλουμε να υπάρξει μία μείωση των κονδυλίων. Από την άλλη, το θεσμικό όργανο Συμβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερε επιδόσει με λιγότερα χρήματα. Αυτή είναι η ουσία και νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται και δεν μπορεί να πετύχει πουθενά σε αυτόν τον κόσμο γιατί τις καλύτερες επιδόσεις πρέπει κανείς να τις πληρώσει. Και τις, ε, δεν βλέπω να συμβάλλουν σε αυτό οι χώρες μέλη. Ε, δεν θέλω να με παρανοήσετε. Ε, ξέρω πολύ καλά ότι πολλές χώρες μέλη έχουν προβλήματα με την προστασία των εξωτερικών του συνόρων και βεβαίως είναι προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρεμπόδιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη ειλικρίνεια σε αυτή τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι έλαβε υπόψη μου τα σώση είπε ο κ. Σφίκελ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πράγματι, οι συμφωνίε που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι καπνοβιομηχανίε, που έχει συνάψει με τι καπνοβιομηχανίε, οδηγούν σε κάποιε πληρωμέ που είναι συνδεδεμένε με ένα στόχο. Δηλαδή θα έπρεπε να συμβάλλουν στην υποστήριξη μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη που μειώνουν το ποστό του λαθρεμπορίου των τσιγάρων. Και πραγματικά θα με ενδιαφέρει κατά πόσο οι χώρες μέλη τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν εισρεύσει σε αυτέ τα έχουν συνδέσει με την επίτευξη αυτού του σκοπού. Γιατί εγώ φοβούμαι πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ πρόκειται για κάποια ποσά που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια και βεβαίω αν κατανεμηθούν στι 27 χώρε 27 χώρες ε, δεν είναι ίσω τόσο αστρονομικά, αλλά παρόλα αυτά ε, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται για παράδειγμα στη Γερμανία από την έκθεση της Όλαφ, ε, πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν γίνει τόσες πολλές, ε, ε, τόσοι, τόσοι πολλές έρευνες της Όλαφ όσο στη Γερμανία σε σχέση με το λαφρεμπόριο τσιγάρων. Είναι το 1 τέταρτο των περιπτώσεων της Όλαφ ασχολούνται στη Γερμανία με αυτό το θέμα. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε όχι μόνο από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίσης και από τη σκοπιά ενός Γερμανού πολιτικού και από τη σκοπιά της Γερμανικής Βουλής, κατά πόσο η Γερμανία τελικά έχει τηρήσει το δικό της κομμάτι της συμφωνίας και τα κονδύλια τα οποία έχουν προέλθει από τις καπνοβιομηχανίες τελικά έχουν χρησιμοποιηθεί και στη Γερμανία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των τσιγάρων. Uh, Θα Ήθελα να προσθέσω μία ερώτηση ε, αναφέρατε ότι βρισκόσατε στη διαδικασία να εξειδικεύσετε τους δείκτες επίδοσης ε, και θα το κάνετε στα τέλη του χρόνου. Τώρα όμως βρισκόμαστε στην ε, διαδικασία συζήτησης του προγράμματος Ηρακλής 3. Δεν έχει γίνει ακόμα για το Ηρακλής 2. Ε, θα ήταν καλό λοιπόν να υπάρξουν οι δείκτες αυτοί για να για το Ηρακλής 2 πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση για το Ηρακλής 3. Και πότε αναμένετε να ολοκληρώσετε την εργασία με αυτούς τους δείκτες. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, αλλά εγώ ίδιος ε, θέλω να υποβάλω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Όλαφ και της Επιτροπής. Εάν κατάλαβα καλά τον κύριο Τσβίκελ, το ελεγκτικό συνέδριο θέτει το ερώτημα ότι δεν έχει νόημα η Όλεφ να διαχειρίζεται ένα δικό της πρόγραμμα, αλλά θα ήταν πιο χρήσιμο η Όλεφ ε, μελλοντικά να περιοριστεί στην καταπολέμηση της απάτης. Ε, νομίζω ότι αυτή ήταν η τοποθέτηση του ελεγκτικού συνεδρίου, εάν κατάλαβα καλά. Και θα με ενδιαφέρει να μας πείτε τι λέτε εσείς κύριε Κάου και η Επιτροπή. Δηλαδή κατά πόσο Μπορούμε να φανταστούμε έναν οργανισμό, ε, μια οργάνωση όπου πραγματικά εφαρμόζεται αυτή η σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Καταρχήν, ε, ο κύριος ε, Κάου θα ήθελα να μας απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας, κυρία Ιβάνοβα, για τα περαιτέρω ερωτήματά σας. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τις ευθύνες της Όλαφ για την οικονομική διαχείριση Ηρακλής 2 και το μελλοντικό Ηρακλής 3 η ειδική έκθεση για την Όλαφ εφαρμόστηκε. Λάβαμε υπόψη και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με διάφορες συστάσεις που έγιναν. Συστάσεις όσον αφορά την ειδική έκθεση για τη διαχείριση της Όλαφ. Αυτή εκδόθηκε το 2011 η ειδική έκθεση. Ο νεο... κ. Γιωβάνι Κέστλερ, ο νεοδιοριστής διευθυντής, μας βελτίωσε τις δυνατότητες της υπηρεσίας όσον αφορά τις έρευνες. Αυξήθηκε το προσωπικό, βελτιώθηκαν οι ερευνητικές διαδικασίες, οπότε σε αυτό το βαθμό λάβαμε υπόψη Τη συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναδιοργανώνεται η υπηρεσία. Ξεκίνησε αναδιοργάνωση από 1η Δευτέρου 2012. Μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τι έρευνες. Ο Γενικός Διευθυντής μας όμως δημιούσε νέα διεύθυνση, υπεύθυνη για πολιτική συμπεριλαμβανομένης τη χρηματοπιστωτικής διαχείρισης. Σαφέστατος ο διαχειρισμός των καθηκόντων από τούδο και στο εξή. Τα πολύ εξειδικευμένα προγράμματα δεν καταργήθηκαν όμως. Στο Ηρακλής 2 και το, και το Ηρακλής 3. Είναι αλληλένδετα. Από την εμπειρία μας αναφέρομαι στο Ηρακλής 2. και αυτά που αποκαμίσαν τι επαφέ με τι δυνάμει τη τάξη στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μας Είδαμε ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που μπορούσαμε να συγχρηματοδοτήσουμε και πού προκυρήθηκαν διαγωνισμοί. και πώς αποκτήσαμε πρόσβαση σε πολύ εξειδικευμένε βάσεις δεδομένων. Δώσαμε πρόσβαση σε αρχές του νόμου διαφόρων κρατών μελών σε πολύ δικευμένε βάσεις δεδομένων. Σας είπα, ο γενικός μας διευθυντής έχει αναδιοργανώσει την υπηρεσία μας ούτως ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση καθηκόντων. Και θέλουμε να θέσουμε και τις προτεραιότητες που συνέστησε το ελεκτικό συνέδριο και προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς εμάς δίνουν προτεραιότητα σε έρευνες, εξωτερικές και εσωτερικές. Όσον αφορά αυτό που είπε η Ιβανόβα για τους δείκτες επιδόσεων. Η Όλεφ πρέπει να δώσει την τελική αξιολόγηση. Θα πρέπει να αφορά το Ηρακλής 2 για την περίοδο 2007-2013. Χρειάζεται τελική αξιολόγηση. Πώς εφαρμόστηκε, πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, τι αποτελέσματα πέτυχε. Το άρθρο 7 της απόφασης αναφέρεται στην τελική αξιολόγηση. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τον καθορισμό δικτών επιδόσεων, πέραν αυτών που έχουμε συμπεριλάβει στην αξιολόγηση συνεπειών και αυτών που εντοπίστηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του 2010. Αυτό είναι ο στόχος μας. Εν τω μεταξύ όμως, όπως προανέφερα, ετοιμαζόμαστε για την απόφαση χρηματοδοτήσεως για το 2013 και θα συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασιών. Με την κοκόλα, την ομάδα εμπειρογνωμόνων που προανέφερα και θα δούμε και πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματά μας. Ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάου. Ε, ίσως να παρακαλέσουμε τον κύριο Ταβέρνα από την Κομισιόν να απαντήσει τις ερωτήσεις που ακόμα κρεμούν. Υποθέτω ότι θέλετε να μου ακούσετε να πω κάτι σχετικά με το ότι χειρίζεται το πρόγραμμα, το ότι χειρίζεται η Όλαφ. Η Όλαφ έχει υβριδικό ε, καθεστω Είναι η υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξήγησε ο συνάδελφο τα μέτρα που ελήφθησαν ούτω ώστε να μην συγχέονται οι δραστηριότητε τη έρευνα και τη ε, πρόθεση προστασία των οικονομικών συμφερόντων μέσω των προγραμμάτων είναι εσωτερική διοργάνωση της, του, φορέα μου. Εκεί δεν έχω σχόλια ιδιαίτερα να κάνω, όμως βέβαια δώσαμε αμέσως αυτό που έθιξε στην γνωμοδότησή του το ελεκτικό συνέδριο, δώσαμε, κάναμε τα δέοντα ε, και για την απαλλαγή. Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω περισσότερα από αυτού του συγκεκριμένου θέματα των διοργανώσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Τσβίκελ να πάρει θέση και να μας πει το πώς αξιολογεί την εφαρμογή των προτάσεών του. Ναι, δεν έχω να προσθέσω πολλά στα όσα ελέγχθησαν, δηλαδή ε, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο θέμα το οποίο αφορά τη διαχείριση του προγράμματος. Διαπιστώσαμε στη γνωμοδότησή μας για το 2011 αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνει όλα. Θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της σε ερευνητικές ε, δραστηριότητες. Ε, το... Παρόλα αυτά, το ελεκτικό συνέδριο σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης εμένει την ε, άποψη ότι η Όλαφ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτό το τομέα της εξαγωγής ερευνών. Ε, ε, αλλά το θέμα είναι κατά πώς θα πρέπει να οργανώνονται τα προγράμματα αυτά, Ηρακλής, 2 ή 3 κλπ. Θα πρέπει να γίνεται αυτό από το ίδιο πρόσωπο ή όχι που κάνει και τις έρευνες. Εμείς θεωρούμε ότι ο διαχειριστής του προγράμματος ίσως δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο πρόσωπο να το κάνει. Τώρα, ε, κάποιες ε, ειδικέ ε, παρατηρήσεις που αφορούν το ποστό συγχρηματοδότησης ή το θέμα της άντλησης περισσότερων πληροφοριών από τις χώρες μέλη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε, ούτως ώστε η Όλεφ να έχει περισσότερες πληροφορίες και στη βάση αυτή θα μπορέσουμε τις ε, ερχόμενες εβδομάδες να οριστικοποιήσουμε την άποψή μας και να τη διαβάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αυτά μόνο μπορώ να πω προς το παρόν. Βεβαίως, ε, όταν διαψώσαμε ότι η συνεδρία θα γινόταν σήμερα, προσπαθήσαμε να επισπεύσουμε τις εργασίες μας και να υποβάλουμε κάποιο σχέδιο. Αλλά παρόλα αυτά περιμένουμε τα οριστικά συμπεράσματα τα οποία θα σας υποβληθούν. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Ο κύριος Μπαλτσίτης θέλει να κάνει μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εδώ και πολλούς μήνες ή χρόνια ε, με πολύ ευγενικό τρόπο εξηγήσαμε οι μεν στους δε, όπως άλλωστε ήδη υπόθηκε εδώ, ε, όσον αφορά αυτή την ε, υβριδικού χαρακτήρα λογοδοσία της Όλαφ, τι μπορεί να γίνει. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει επιτέλους να λυθεί. Και συμφωνώ με το ότι η Όλαφ δεν είναι δυνατόν να αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή του προγράμματος, αλλά θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στις ανακρίσεις, στις έρευνες και ε, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα πάνε όλα στη θέση τους και δεν θα σπαταλήσουμε το χρόνο για να εξηγούμε πράγματα τα οποία συζητούμε εδώ και πολλούς μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή ήταν μια πολιτική αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Ιβάνοβα να πάρει το λόγο καταλεκτικά και στη συνέχεια να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ κυρία Ιβάνοβα. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σχετικά με το ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες πολέμησης ε, του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Θέλουμε όμω και ε, μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερο συντονισμό, καλύτερη κατανόηση σε σχέση με τη δράση των κρατών μελών αφενό και τη Επιτροπή Αφετέρου. Σε αυτό το στάδιο θα προετοιμάσουμε δεύτερο έγγραφο εργασίας για τα βασικότερα και δυσκολότερα ζητήματα και θα συμπεριλαμβάνει πιθανές λύσεις για το μέλλον και όπως είπε και ο κύριος Τουίκελ του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούσαμε να συντονιστούμε όταν είναι έτοιμο δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του θα μπορούσαμε να επιφεληθούμε για να παρουσιάσουμε και εμείς το δεύτερο έγγραφο εργασίας Ιδού Πρόεδρε και σταματώ εδώ. Ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστούμε επίσης πολύ τον κύριο Κάου, τον κύριο Ταβέρν και τον κύριο Τσβίκελ για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί και ως Κοινοβούλιο ως προς το θέμα αυτό, όπως και για άλλα θέματα, θα θέλαμε να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα εν σχέση με το τι κάνουν οι χώρες μέλη. Αυτό είναι ένα βασικό θεσμικό πρόβλημα και ελπίζουμε στο πλαίσιο της ε, περαιτέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης θα βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τα κοινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εδώ έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας του, της Επιτροπής Προπολογισμών και εμείς ε, θα γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα της κυρίας Ιβάνοβα και εδώ είναι η συγγήτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναλάβατε τόσο πολλές ευθύνες. Σας δίνω το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ. Τελευταία φορά με ακούτε, το υπόσχομαι. Λοιπόν, για τα διεθνή εργαλεία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ανακοίνωση 662 του 2011 ότι θα πρέπει να αναλάβει λένε και σημαντικότερο ρόλο αυτή η χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 και άρα είναι εξαιρετικά επίκαιρη και χρήσιμη η έκθεση αυτή. Αναπτύχθηκαν ε, πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορα νέα εργαλεία χρηματοδότησης. Αν δούμε τις λεπτομέρειες θα συνειδητοποιήσουμε ότι τέτοιου είδους εργαλεία ε, υπάρχουν και σε άλλους τομείς, έρευνα και ανάπτυξη, γεωργία κτλ το κυλιόμενος χαρακτήρας του, δηλαδή ε, ο αναπληρούμενος χαρακτήρας του ταμείου αυτού επιτρέπει μεγαλύτερη μόχλευση. Αυτή είναι η διαφορά. Ε, ας περάσω τώρα στην ε, άποψη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για αυτά τα εργαλεία. Μέσα στην γνωμοδότησή μου τονίζω διάφορα σημεία όπως π.χ ο ορισμός ε, των εργαλείων αυτών, των μέσων αυτών, ε, μέσα ε, στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο οι νέες διατάξεις σε, σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ορισμό σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, ε, τα κενά χρηματοδότησης ε, πρέπει να καλυφθούν για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ε, δημόσιο χρήμα. Αλλιώς θα προκύψουν στρεβλώσεις στην αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Υπάρχουν δύο σχόλια. Πρώτον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή τους και τη χρηματοδότηση, το δεύτερο σκέλος, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΤΠΑ. Τονίζω, βασιζόμενοι στι παρατηρήσει του ελεγκτικού συνεδρίου, ότι θα πρέπει όντω να δοθεί μια λύση προτού αυξηθεί ο αριθμό των νέων χρηματοδοτικών μέσων στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αποφάσισα να υποβάλω και σχετικέ τροπολογίε. Τροπολογίες ε, που ουσιαστικά είναι συστάσεις και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε προτού πολλαπλασιάσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Χρειαζόμαστε καλύτερα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, παραδείγματο χάρη, χάρη στα οποία θα έχουμε ε, συγκεκριμένους ε, και αποτελεσματικούς δείκτες που θα βασίζονται ε, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους στόχους για να μπορούμε στη συνέχεια να αποτιμούμε την αποτελεσματικότητα των νέων χρηματοδοτικών μέσων. Θα ήθελα να απευθύνω, αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε, κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, έχει την πρόθεση η Επιτροπή να μας ενημερώσει μέσω έκθεσης ή ανακοίνωσης για τη χαρτογράφηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που λειτουργούν με κονδύλια του προπολογισμού της Ένωσης ε, στα πλαίσια του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερον, τα μέσα που αναπτύσσει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύουν τους ίδιους ή σχεδόν τους ίδιους δικαιούχους ε, σε κάποια προγράμματα ε, των διαρθρωτικών ταμείων ε, και προγράμματα για την έρευνα ε, και την ανάπτυξη. Αποδέκτες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Με ποιο τρόπο θα αποφύγει την επικάλυψη ανάμεσα στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον θα αυξηθεί ο αριθμό των ταμείων. Ευχαριστούμε. Χαιρετίζω και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλατε κι εσείς να τοποθετηθείτε για να μας διευκολύνετε για τη συνέχεια της συζήτησης, παρακαλώ ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Με τα χαράς μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή και την εισηγήτρια για τη σημαντική συμβολή της. Θα πιαστώ από το τελευταίο σχόλιο της εισηγήτριας για να αρχίσω την παρουσίασή μου. Στο τωρινό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όντως υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και κάποια από αυτά παρουσιάζουν τέτοιους κινδύνους επικάλυψης και φυσικά έχει επίγνωση αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και σκοπεύουμε να ε, διαχειριστούμε αυτούς τους ε, κινδύνους επικάλυψης, οι οποίοι οφείλονται σε ανεπαρκή συντονισμό. Προτείνουμε ένα μικρότερο λοιπόν αριθμό χρηματοδοτικών μέσων με σαφότερα σημεία διεπαφής για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των προγραμμάτων όπως τα προγράμματα SIP το 2020 προτείνουμε αυτό συγκεκριμένα για την περίοδο μέχρι το 2020 προτείνουμε μικρότερο αριθμό μέσων με καλύτερες διεπαφές. Επίσης, οι προτάσεις μας βασίζονται στις παρελθούσες εμπειρίες με στόχο να ε, ε, υπάρχουν ισότιμοι όροι και να αποφύγουμε το shopping ε, ε, την ε, επιδίωξη την να χρησιμοποιήσει κανείς το πλέον προσοδοφόρο χρηματοδοτικό μέσο. Κάποια κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια χρηματοδοτικά μέσα παρότι επικαλύπτονται με υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα άλλων τομέων. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτά τα κράτη-μέλη. Για να το αποφύγουμε όμως, ε, στα διαρθρωτικά ταμεία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο πλαίσιο, βάσει του οποίου θα υπάρχει δυνατότητα ε, μικτής χρήσης χρηματοδοτικών μέσων οι χώρες, ε, οι περιοχές, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν βάσει των νέων διατάξεων να συνδυάσουν ε, χρηματοδότηση από διάφορα μέσα με στόχο την επίτευξη σαφών στόχων σε κάθε τομέα πολιτικής. Αυτή είναι η λύση μας, η ενοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων και ο προσδιορισμός ε, ισχυρών κινήτρων για την χρηματοδότηση στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων. Ο συνδυασμός των δύο θα μας δώσει την απάντηση κατά τη γνώμη μας. Τώρα, Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις από βουλευτές του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα και η ίδια η Επιτροπή έκανε μια ανασκόπηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Βεβαίως στη διάθεσή σας είμαστε, αν χρειάζεται κάτι άλλο μπορούμε να σας δώσουμε τις σχετικές πληροφορίες. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτό το σχέδιο γνωμοδότης, κυρία Σιβάνοβα. Το καλωσορίζουμε διότι αποδίδεται το βάρος ε, στην, ε, στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της ε, ταυτόχρονης χρήσης διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αποτελεσματική χρήση αυτών. Όλα Όλοι αυτοί ε, που εμπλέκονται στην αλυσίδα για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα εντάσσονται σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διέπει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα. Σε σχέση τώρα με τι δωρεέ, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και τεχνική πραγματογνωμοσύνη από όλου αυτού ε, του φορεί. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και για χρηματοδοτική πραγματογνωμοσύνη. Όπω σωστά είπατε, είναι αλληλοσυμπληρούμενα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Θεωρούμε όντω ότι τα μέσα αυτά δεν συνιστούν κρατική παρέμβαση, δημόσια παρέμβαση. Έχουμε την εντύπωση ότι η εξάντε αξιολόγηση για τις ενισχύσεις ανά ανάχρηματοδοτικό μέσο είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να επιτύχουμε τους στόχους ανά τομέα πολιτικής. Στα πλαίσια κάποιων ελέγχων, κυρίως στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων, είχαμε κάποια ευρήματα που αποκαλύπτουν ε, κινδύνους αλληλεπικάλυψης. Ε, Ο κίνδυνο δεν είναι εγγενή στα χρηματοδοτικά μέσα, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται σε αναπερίσταση τα χρηματοδοτικά μέσα. Οι όροι εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων προσδιορίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν μιλάμε για το τομέα της συνοχής ισχύουν διαφορετικά κριτήρια σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με άλλους τομείς. Ας πάρουμε τον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με την εφαρμογή είναι όντως ίσως υψηλότερος λόγω του αριθμού ε, των στρεμάτων, των εκταρίων και λόγω των περίπλοκων κανόνων ε, που καλούνται να εφαρμόσουν οι διαχειριστικές αρχές. Επίσης, ε, αναπτυξιακά προγράμματα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Και εκεί υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος. Όντω υπάρχουν τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις και επεξεργαζόμαστε ένα καταλληλότερο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτούς τους τομείς. Όμως, προσοχή, υπάρχει το θέμα του κινδύνου και της απόδοσης, κάτι που ισχύει για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και στον τομέα σύνοχης, αλλά δεν πρέπει να ε, βλέπουμε μόνο τις διαφορές ε, και να μην συνειδητοποιούμε και τις διαφορές που ισχύουν τους ή σε κάθε αγορά. Προτού αποφασίσουμε, πάρουμε αποφάσεις ε, για την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, πρέπει πρώτα να ορίσουμε το κενό χρηματοδότησης, ε, ε, να λάβουμε υπόψη τις επενδυτικές ανάγκες ε, της αγοράς, της, τη μη ικανοποιητική κατάσταση ως προς επενδύσεις, ανατομέα κτλ. Δηλαδή απαραίτητα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν αυτά τα κενά χρηματοδότησης γιατί δεν είναι στατικά, μετεξελίσσονται ανά τομέα, γεωγραφική περιοχή, παραδείγματο χάρη και άρα κατά τη γνώμη μας δεν γίνεται με αξιόπιστο τρόπο να ποσοτικοποιήσουμε αυτά τα κενά. Ούτως ή άλλως δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε για το 2013 ε, ε, ενώ το χρηματοδοτικό μέσο ε, έχει κύκλο ζωής 10 ή 20 χρόνια. Για να αποφύγουμε τις τρευλώσεις στην αγορά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τα χρηματοδοτικά μέσα αλλά και για τις δωρεές που ε, ορισμένες φορές ε, προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη στρέβλωση. Για να περάσω τώρα στις διάφορες εκθέσεις, ε, τις διάφορες ελεγκτικές εκθέσεις και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, τα ΣΥΠ. Οι συστάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν οριζόντια, αλλά συμφωνήθηκε με το συνέδριο ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις για το επόμενο πολιετές πλαίσιο, γιατί σχετίζονται μάλλον με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό και άρα ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάλι για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τις συστάσεις και για το τωρινό πλαίσιο βάσει της ανακοίνωσης ε, της Επιτροπής του Φεβρουαρίου του 2011 και θα να υπόψη και για ε, την εκπόνηση του επομένου πλαισίου διότι οι κοινοί κανόνες για το στρατηγικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνουν ε, ξεκάθαρους κανόνες, ε, σαφέστερους κανόνες ε, για τα χρηματοδοτικά μέσα στην ε, τωρινή προγραμματική περίοδο έχουμε συλλέξει διάφορες ε, βέλτιστες εμπειρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την εκπόνηση του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου. Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι Σύμφωνοι μου απολύτω ε, με τη θέση τη εισηγήτρια ότι η συμβολή των χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Εδώ και 15 χρόνια χρησιμοποιούνται. Ε, έχουν αξιολογηθεί σε επίπεδο Επιτροπής κράτους μέλους, στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Έχουμε ήδη εντοπίσει κάποια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ασχολούμαστε με αυτά. Πάντως με κάποιες ε, προσαρμογές ε, θα μπορούσαν να έχουν ένα πιο πάγιο ρόλο τα χρηματοδοτικά μέσα στις διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ε, γνωρίζετε όλοι ότι είναι περιορισμένα τα μέσα που τους αποδίδονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Χατζημαρκάκης θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, είπατε, είναι το πρόβλημα. Και πράγματι η εφαρμογή γίνεται στις χώρες μέλη. Και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς εδώ και το οποίο είπε και η κυρία Ιβάνοβα, ε, κυρίως στο σημείο 2 του σχολείου, ότι μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομικός ορισμός και ότι η χρησιμοποίηση από τις χώρες μέλη ε, ε, γίνεται με ένα εξατομικευμένο τρόπο, αν θέλετε, και συνδέεται με υψηλού κινδύνου. Τώρα, η κατάσταση έχει ω εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερω, ε, χρησιμοποιεί τη δική της ε, τράπεζα για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτά τα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι ε, το European Investment Facility εν μέρη ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που το κάνουν. Αλλά εγώ δεν το άκουσα να αναφέρεται εδώ. Και θυμάμαι ότι είχαμε μια σύντηση με τον συνάδελφο κύριο Γκάιερ ε, και οργανώσαμε κάποιες συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε κάποια πράγματα από τις εμπειρίες της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας ε, όσον αφορά τη χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών μέσων για να αναπτύξουμε κάποιο μοντέλο. Ε, και εσείς αναφερθήκατε σε κοινέ προδιαγραφές άλλωστε ένα κοινό πρότυπο, αν θέλετε, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις χώρες μέλη. Εσείς ε, μιλήσατε για ε, μια εκούσια χρησιμοποίηση και εγώ διαρτώμαι κατά πόσο δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή. Αλλά εάν ε, δεν γίνει αυτό, διατρέχουμε σημαντικούς κινδύνους. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το διατυπώσουμε κάπως πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, αυτό το πρότυπο το οποίο έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί πράγματι να, να πρέπει πράγματι να εφαρμόζεται ε, και στις χώρες γιατί υπάρχουν τώρα κάποια χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είναι της μόδας και αν αφήσουμε μεγάλο περιθώριο ελευθερία χώρε μέλη θα αυξηθούν οι κίνδυνοι. Ο κύριος Γκάιερ θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ο Γιώργος ε, έφυξε κάποια θέματα τα οποία ήθελα και εγώ να θέσω. Πράγματι, τα χρηματοδοτικά μέσα ε, είναι κάτι, εφόσον χρησιμοποιούνται έτσι αυθαίρετα, είναι κάτι σαν μαγικά όπλα. Πρώτον, τα χρηματοδοτικά μέσα ε, μπορούν να εκπληρώσουν την, ε, τις εξαγγελίες τους ε, για να προσεγγίσουν περισσότερο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχουμε. Και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην τελευταία του έκθεση είπε ότι αυτού του είδους ε, χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού με τον οποίο για τον οποίο διαβουλευόμεθα με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Κάτι που ανέφερε ήδη και η κυρία Ιβάνοβα στη δική της γνωμοδότηση, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Αλλά δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Και η ανησυχία μου είναι ότι εάν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, να οριστεί δηλαδή το νομικό πλαίσιο για τα χρηματοδοτικά μέσα, τότε τα μέσα αυτά θα συνένονται με πολλούς κινδύνους και πραγματικά ανησυχούμε. Συνολικά συμπλέουμε με τη γραμμή της εισηγήτριας, αλλά θα θέλαμε στο σημείο υπαρθμό 3 να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη διατύπωση όσον αφορά τους κινδύνους της αποτυχίας της αγοράς και των ε, κενών χρηματοδότησης. Και στο σημείο υπαριθμών 7, και ταιριάζει αυτό με τα όσα είπα προηγουμένω, να διατυπωθεί πιο ξεκάθαρα ότι μια ανάμειξη των χρηματοδοτικών ε, μέσων τελικά αυξάνονται οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά. Τώρα, στην έκθεση απαλλαγής το ζητήσαμε ήδη και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και πιστεύω, Γιώργο, αυτό ταιριάζει με τη δική σου αντίληψη για αυτό το πρότυπο, αυτή τη μήτρα, εάν θέλεις, ε, ε, προδιαγραφών. Θα πρέπει να μερμήσουμε να υπάρξει μια πολύ ε, ρεκτική παρακολούθηση των κινδύνων ούτως ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις εισφορές τους εάν θα πρέπει η τράπεζα αυτή να χρηματοδοτήσει περαιτέρω μέσα. Αλλά θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο πού προέρχονται στην περίπτωση αυτή τα κονδύλια. Και εμείς θα θέλαμε να υπάρξουν εδώ κάποιες κόκκινες γραμμές. Δηλαδή να υπάρξει μια ξεκάθαρη άποψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού στην έκθεση πρωτοβουλίας, δηλαδή να αποκλείονται οι κερδοσκοπίες στην αγορά μέσω τέτοιου είδους χρηματοδοτικών μέσων και να μην ε, εκπονούνται από κοινού ε, με κάποιες ε, τράπεζες ή οργανισμούς που έχουν τη βασική τους έδρα σε φορολογικούς παραδείσους κατά την άποψή μας ε, κάτι τέτοιο δεν θα ζημίωνε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Αντιθέτως. Ευχαριστούμε <coughs> πολύ και τώρα θα, θέλαμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα πριν τοποθετηθεί η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και που ανέχθηκαν όλη μέρα την παρέα μας και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή της ε, και αυτά είναι όλα όσα έχω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Ε, ίσως ε, θα μπορούσατε να τοποθετηθείτε στα θέματα που αναφέρθηκαν, τα ερωτήματα όσον αφορά την διευκρίνηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επεκταθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτα κοινή ορισμή. Δεύτερον, για τους φορείς που εμπιστευόμαστε, για να χρησιμοποιήσουμε την ε, έννοια που χρησιμοποιεί ο δημοσιονομικός κανονισμός. Και μετά οι μήτρε και κόκκινε γραμμέ. μετά. Η αύξηση του κεφαλαίου να πηγαίνει κάπως μακριά, αλλά μπορώ να πω κάποιε κουβέντες και γι' αυτό. Ορισμοί. Στο δημοσιονομικό κανονισμό έχουμε κοινό ορισμό που θα είναι υποχρεωτικός και για τα χρηματοδοτικά μέσα και για τα διεθνωτικά ταμεία. Διότι στα πλαίσια των κοινών διατάξεων των διεθνωτικών ταμείων ο ίδιος ορισμός χρησιμοποιήθηκε και αντεγράφει στο πλαίσιο. Όλα τα δημοσιοτικά μέσα, τα συγκεκριμένα, τα ειδικά που προτείναμε, παραπέμπουν στο δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά τους ορισμούς και γι' αυτό θα εφαρμόζουν όλοι αυτό τον ορισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά πέραν αυτού. Δεν ορίζουμε μόνο τα χρηματοστικά μέσα και τα προϊόντα, αλλά θέλουμε να έχουμε συνεπή ορισμό για βασικές έννοιες όπως ε, συνέπεια πολλαπλασιαστική, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διότι βλέπουμε πολλαπλές ερμηνείες γι' αυτό και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι στην έκθεσή μα, στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να χρησιμοποιούμε συνεχώ τι ίδιε έννοιε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια έννοια. Όσον αφορά το πλαίσιο, πολλή προσοχή έχει δοθεί στην παράλληλη εξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού και των κατεξισοδότηση πράξεων που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο τον Μάιο. Αυτό από τη μια και απ' την άλλη κοινέ διατάξει εθνοτικά ταμεία και κατεξουσιοδότηση πράξη. Και όπου είναι δυνατόν θέλουμε να υπάρχει συνέπεια και συνοχή. Υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν ανάγκες διαφορών. Δεν πάντα γράψουμε τα πάντα. Όπου είναι δυνατόν θέλουμε να θυγραμμίσουμε να το πλαίσιο. Τα θετικά ταμεία, το πλαίσιο θα είναι πληρέστερο, εκ των προτέρων καθορισμένο, με σαφείς κανόνες από την πρώτη μέρα δεν θα γίνουν ρυθμίσεις εκ των υστέρων. Τώρα, για τις αξιόπιστες, τους αξιόπιστους φορείς. Μπορεί να χειριστεί και να εφαρμόσει τον προπολογισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άμεση διαχείριση, στον τομέα όμως των χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτό εφαρμόζεται έμεσα και είναι συνηθισμένο, εμπιστευόμεθα τρίτα μέρη. Και αυτή είναι η, αυτή είναι έμπιστη Σε ποιους μπορούμε να αναθέσουμε την εκτέλεση του προπολογισμού και ποιος θεωρείται ως έμπιστος φορέας περιγράφεται στο δημοσιονομικό κανονισμό για την επόμενη περίοδο. Είναι πολύ περιορισμένο αριθμός. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδομήσεως και Ανάπτυξης, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Συμβούλιο της Ευρώπης και Τράπεζα, διεθνή Χρηματοπιστωτική Φορή και εθνικέ τράπεζε και Ιδιωτική Φορή με δημόσια αποστολή. Όχι όμως ιδιωτικό χειριστή ταμείου ούτε ιδιωτική τράπεζα. Αυτή δεν είναι έμπιστη φορείς. Άρα αυτό προβλέπεται ήδη σαφώς στο δημοσιονομικό κανονισμό. Επιπλέον υπάρχουν απαιτήσει σχετικά με την επιλογή αυτών. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νικόδοση Απαντήσεω, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πρέπει να αναφέρονται ρητά σε πράξη συγκεκριμένη. Αν δεν αναφέρονται, πρέπει να εφαρμόζεται μια δίκαιη διαφανή διαδικασία και κανόνες επιλογής. Όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να περάσουν μια αξιολόγηση μέσω έξι πυλώνων εκ των προτέρων, ούτω ώστε να έχουν διαδικασίες που να αντιστοιχούν σε αυτές που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, για τις μήτρες υπάρχουν δύο επίπεδα επεξεργασίας αυτών. Πρώτον, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασαν όλα τα χρηματοστικά μέσα σε, στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου και τα μαθήματα που πήραμε και καταλήξαμε σε κανόνε που θέλουμε να προωθήσουμε στο μέλλον και θέλουμε να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο. Αυτή ήταν η βάση τη προτάσεώ μα όσον αφορά του δημοσιονομικού κανονισμού στη συζήτηση με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι κανόνες θα υποβληθούν τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τις κατεξουσιδότηση πράξης, βάσει των ίδιων εμπειριών και θέλουμε να έχουμε κανόνες υποχρεωτικούς, θα πρέπει να τηρούνται από όλες τις υπηρεσίες εν τη εκτελέση το, των ε, χρηματοπιστωτικών μέσων και για τα διεθνωτικά ταμεία. Και τρίτη ομάδα θα εφαρμόζεται μόνο για μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή όπου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλλει στι υπηρεσίε τι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά πιο τεχνικά ζητήματα που είναι αποτέλεσμα αξιολογήσεως των εμπειριών μας. Διαφορετικά ταμεία. Διαφορετική κατάσταση. Πρέπει να ορίσουμε εκ των προτέρων όλους τους κανόνες, διότι οι χειριστικέ αρχές αποφασίζουν εκ των υστέρων πώς θα το κάνουν αυτό. Πρέπει να συμμορφωθούν όμως με τους κανόνες. Τι θα κάνουμε εδώ. Θα δώσουμε δύο ε, μορφές συμπληρωματικών παρεμβάσεων έκτακτα μέτρα, αυτό που ανέφερε ο κύριος Χατζημαρχάκης, off the shelf, όπως αποκαλείται αγγλιστή, έτοιμα χρηματοστικά μέσα σε διάφορους τομείς πολιτικής. Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να τα πάρουν αυτά τα μέσα. Υπάρχει προέγκριση όσον αφορά τις αναφορές, το σχεδιασμό και συμμόρφωση με κρατικές ενισχύσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη καινοτομία και περαιτέρω προσαρμογή μετά και κοινά μέσα μετά που ακολουθούν του κανόνε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Άρα θα υπάρχει μια μήτρα, ένα πρότυπο. Κανόνε Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά η συμμετοχή θα είναι θελοντική. Τρίτον, αυτό που έχουμε τώρα στο MFF. Οι διαχειριστικέ αρχέ αποφασίζουν για τα δικά τους μέσα. Όμως πρέπει να συμμορφώνονται με κοινέ διατάξει και κατεξουσιοδότηση πράξη και εφαρμοστικού κανόνε. Οι κόκκινες γραμμές. Συμφωνούμε όσον αφορά την οικονομική αντιμετώπιση και την ανάγκη επαρκών διατάξεων για να αποφευθεί φοροδιαφυγή. Και τα βάλαμε όλα αυτά στο δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν είναι μια της απαιτήσει αυτού του κανονισμού αλλά θα γίνουν διευκρινήσεις στις κατεξουδότητες συμπράξεις. Όχι μόνο στις έμπιστους φορείς θα ισχύει, αλλά στους πάντες. Πρέπει να εφαρμόζονται τους κανόνες στις συμβάσεις τους με μεσάζοντες. Για την κεφαλουχική αύξηση, αύξηση κεφαλαίου, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμηση και Επενδύσεων δεν πρέπει να πω για την πολιτική χρειά, αλλά τα χρηματοστικά μέσα συνεπάγονται μοίρασμα των κινδύνων με του διάφορου εμπλεκόμενου φορεί και άρα επηρεάζουν την επάρκεια κεφαλαίων των διαφόρων θεσμικών οργάνων και τη ρευστότητά τους. Συνεπώς, για την ώρα μεν μπορούμε να αυξήσουμε τα κοινά μέσα και τα μέσα κοινή αντιμετώπιση των κινδύνων, αλλά σε κάποια φάση θα πέσουν πάνω σε έναν τοίχο. Είτε θα πάρει περισσότερο κεφάλαιο, οι άλλε μορφέ στήριξη η Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεω και Ανοικοδόμηση, δεν μπορεί να επεκταθεί όσον αφορά την χρήση κοινών μέσων. Άρα υποστηρίζω τη δήλωση των μελών της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Έχουμε μια ψηφοφορία οι τροπολογίε θα πρέπει να κατεθούν μέχρι τις 3 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι και στις 21 Μαΐου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Εδώ λοιπόν περατώναν τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περάμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για, το, για έναν κανονισμό της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Συντάκτης της έκθεσης είναι ο κύριος Γκάιερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους εναπομείναντες συναδέλφους για την υπομονή τους. Υπάρχει ένα νέο μας προτείνει η Επιτροπή για το οποίο θα επιθυμούσα τον τίτλο «Κοινωνική πρόοδος και κοινοτομία» και όχι «Κοινωνική αλλαγή» για να γίνει ξεκάθαρο ποια κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσει. Λοιπόν, κατάλαβα ότι εδώ το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα επιπλέον εργαλείο στο τομέα της πολιτικής απασχόλησης ε, πέρα από τα όρια του EFSF που να προβλέπει νέες ε, πρακτικές και νέα εργαλεία και να τα δοκιμάζει πειραματικά μάλλον, να χρηματοδοτεί την ε, δοκιμή τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ευρώπη 2020 και κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας. Εγώ τήρησα πολύ αυστηρά, προσπάθησα να τηρήσω αυστηρά τα, ως ορίζοντας καθήκον της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Αλλά δεν μπόρεσα να μην προτείνω κάποιες αλλαγές, γιατί στο βαθμό που στατεύουν σε υπόθεση της ευρωπαϊκής πολιτικής, προσκρούσε μία τρόπο δεινά ηρωνική αντίφαση μεταξύ των στόχων που θέλουν να επιτύχουν αυτά τα προγράμματα και όπως φαντάζεται κανείς σε ένα χώρο 27 χωρών και πολιτών που πρόκειται να υποφεληθούν αυτά τα προγράμματα και τελικά έχουμε ένα πολύ ισχνό, πενιχρό ποσό το οποίο λόγω ακριβώς του περιορισμού του δεν είναι δυνατόν να χρησιμεύσει για την επίτευξη των στόχων. Και αυτή δεν είναι κριτική για την Επιτροπή, αλλά θα ήθελα στην ίδια τη διατύπωση να σε επισημάνω ότι εδώ έχουμε πολύ περιορισμένα μέσα στη διάθεσή μας, άρα έχουμε περιορισμένες ε, παρεμβάσεις στο πλαίσιο ορισμένων προγραμμάτων καινοτόμων. Γι' αυτό λοιπόν τόνισε επίσης ότι τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν υποδειγματικό χαρακτήρα και θα πρέπει να επιφέρουν μια σαφώς αναγνωρίσιμη προστιθέμενη αξία. Και αυτό με δημιουργεί κάποιε ανησυχίε γιατί και αυτό είναι το δεύτερο μαγικό όπλο όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων εκ μέρου τη Επιτροπής κατά την ε, προπαρασκευή τη Ρύθμιση των διαφόρων τομέων στο πλαίσιο του επόμενου πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου να υπάρχουν δηλαδή συνέργειε μεταξύ των διαφόρων ταμείων και μεταξύ των διαφόρων προγράμματο. Εμεί όμω είμαστε ελεγκτέ του προπολογισμού και το ζήτημα τη συνέργεια, ναι, μεν είναι χρήσιμο, αλλά εκεί που υπάρχουν επικαλύψει και αποκτούν ένα αφαίρετο χαρακτήρα, τα πράγματα δυσχεραίνονται εξαιρετικά. Γιατί θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι είναι στο πρόγραμμα που του προσδίδει ένα χαρακτήρα να μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες όπου τα ίδια ε, εργαλεία, τα ίδια προγράμματα μπορούν να δημιουργηθούν από δύο εργαλεία, ε, δημιουργούμε επικαλύψεις και ασάφειες στον προγραμματισμό. Και δεν πρόκειται για αληθινές ε, συνέργειες. δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους συνέργειες μπορούν να υπάρξουν εδώ πέρα. Και δημιουργούμε, και τουλάχιστον αυτή είναι η ανησυχία μου, μια κατάσταση όπου σε τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θα έρθει και θα μας πει ότι είναι εντελώς ασαφές ποια προγράμματα θα πρέπει να χρηματοθούν από το ΙΦΣΕΦ e και ποια από αυτό το πρόγραμμα. Ε, και ίσως σε μια χώρα θα έχουμε χρηματοδότηση από το ΙΦΣΕΦ e και σε, ένα άλλο, σε μια άλλη χώρα θα χρηματοδοθούν αυτό το πρόγραμμα. Και τα πράγματα θα δυσχερανθούν πάρα πολύ, όταν συμβεί κάτι τέτοιο και τελικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ίδιο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ίδιο το πρόγραμμα και από την άλλη από το EFSF, τη μια από το ένα και την άλλη από το άλλο. Ε, το οποίο e FSF τελικά θα χρηματοδοτείται μόνο από την Επιτροπή. Δηλαδή, ορισμό, η έννοια της συνέργειας δεν μας εξυπηρετεί και τελικά οδηγεί σε μεθοδολογικές επικαλύψεις και επικαλύψεις όσον αφορά το περιεχόμενο της χρηματοδότησης. Γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της συνέργειας. Επιφυλάσσεται λοιπόν η Επιτροπή να ορίσει τους τομείς στόχων που έχει σαν σκοπό να καλύψει το πρόγραμμα αυτό ε, τουλάχιστον αφορά τα εκάστοτε ποσοστά με αυτούς τους τρεις σκοπούς που πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, και υπάρχει δυνατότητα ποσοστίας αλλαγής. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει πιο σαφής οριοθέτηση γιατί εδώ μπορούν ενδεχομένως να υπάρχουν πολιτικές ε, προτεραιότητες και διάφορες, ε, που να προκύπτουν διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες από το Συμβούλιο και αναλόγως να χρησιμοποιούνται τα κάστα εργαλεία για να εκπληρώνουν τις πολιτικές σκοπιμότητες του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα ήταν καλό να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη οριοθέτηση και θεωρώ ότι θα ήταν πιο εφεκταίο αν είχαμε κατέτος ε, παρακολούθηση και εάν η Επιτροπή μπορούσε να αποφασίσει ε, να γίνεται αυτό ετήσια και όχι κάθε δύο χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Κριστίνα Αστούριας από την Επιτροπή. Κυρία Αστούριας, ε, θέλετε να τοποθετηθείτε για... σε σχέση με τα θέματα που έθεσε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Θα τα πω γρήγορα γιατί είναι 6 παρά 20 σε σχέση με την επικάλυψη των προγραμμάτων του, Ευρω... του και ε, ΣΥΠ από την άλλη. Θα σε ευχαριστώ που μου κάνατε αυτή την ερώτηση διότι το είχα θέσει και στην αρχή του προγραμματισμού. Είναι σαφέστατη η απάντηση. Είναι αλληλοσυμπληρούμενα αυτά τα προγράμματα και αναφέρεται στο άρθρο 8 της πρότασης κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, συντονίζει προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ τα ΣΥΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη έχουν μάλλον ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή θα έλεγα διάσταση. Οπότε δεν γίνεται, δεν είναι εφικτή η επικάλυψη. Ζητήσατε συγκεκριμένα παραδείγματα για τα προγράμματα. Ναι, πρόκειται για ε, δραστηριότητες ανάλυσης, στατιστικών στοιχείων, ε, η διάδοση κοινών ε, μεθόδων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τα ΣΥΠ και όχι το ΕΚΤ. Τα κονδύλια τώρα. Διαβάστε για τα δύο προγράμματα Progress την έκθεση ενδιάμεση αναθεώρησης. Ε, θα τη δώσουμε στη γραμματεία της Επιτροπής. Προκύπτει ότι το πρόγραμμα Progress είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα με κονδύλια αντίστοιχο, όπως και για το ΣΥΠ. εν γέννη παρατηρείται προστιθέμενη αξία και η, διαχείριση σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο δεν παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Αυτά φαίνονται όλα μέσα στην ενδιάμεση έκθεση. Σε σχέση με τα ποσοστά, προτείνουμε τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην τωρινή κατάσταση. Για τα πρόγκρες προτείνουμε αύξηση 9%. Αλλά δεν ισχύει αυτό για τα προγράμματα καινοτομία, τα λεγόμενα SIP. Ja, vielen Dank, Frau Asturias. Damit können wir den Punkt abschließen. Es sei denn, der Herr Geier möchte noch mal... Ο κύριο Γκάιερ ίσω θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Εάν όχι, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, το σημείο υπαριθμών 13 που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Και εδώ η συγκεκριτή είναι ο κύριο Χατζημαρκάκης. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε το 2006. Ήταν μια συνέπεια της αντιευρωπαϊκής ατμόσφαιρας σε ορισμένες χώρες μέλη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στη Γαλλία μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και τότε η Επιτροπή θεώρησε ότι μπορεί μέσω αυτού του Ταμείου να, αντιστρέψει, να αναστρέψει το κλίμα. Και υπήρχαν ορισμένοι βουλευτές εδώ, ορισμένε ομάδες που το έβλεπαν αυτό ιδιαιτέρως κριτικά γιατί το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν πανάκια. Στο ταμείο αυτό ε, υπάρχουν 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυτά είναι απομεινάρια κυρίως από το Ταμείο Γεωργίας και αυτό είναι ο λόγος που η Επιτροπή Γεωργίας ε, έχει λόγο εδώ, καθώς και η Επιτροπή Κοινωνικών ε, Υποθέσεων. Τώρα, το μεγαλύτερο ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί ήταν 133 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτό δείχνει ότι η προθυμία να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζήτημα της επιμόρφωσης και πραγματικά αυτό θα πρέπει να το χαιρετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Και επειδή δεν υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια ή επειδή τα κριτήρια δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρα το έτος της ίδρυσης του Ταμείου το 2006, το 2009 ορίστηκαν κάπως πιο επακριβώς. Και τώρα βρισκόμαστε στο γύρο αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων και εδώ πρόκειται για τις τροπολογίες στην έκθεση την οποία θέλω να σας παρουσιάσω και πρόκειται για 12 συνολικά τροπολογίες. Ε, ξέρω ότι η συνάδελφος Όρτης πρόκειται να κάνει ε, άμεσα κάποιες προτάσεις. Η πρώτη τροπολογία αφορά τη συγχρηματοδότηση. Μέχρι τώρα ήταν 50% το ποστό συγχρηματοδότησης και τώρα ε, θα πρέπει να αυξηθεί στο 65% αλλά εφόσον υπάρχουν ξεκάθαρα επακριβώς ορισμένα κριτήρια για την αύξηση της χρηματοδότησης όσον αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Επίση, θέλουμε να βοηθήσουμε τους, ε, να συμπεριλάβουμε μάλλον του καλλιεργητέ και τους ε, ε, ελεύθερους επαγγελματίες και πραγματικά είναι μια ορφή απόφαση γιατί και οι χωρικοί και οι γεωργοί και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες μπορούν να επιφολούν αυτό το ταμείο ή πλήττονται από την κρίση. Ε, η κρίση θα πρέπει επίσης να ήταν ένα κριτήριο για κινητοποίηση των κονδυλίων θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια διασύνδεση με την χρηματοπιστωτική κρίση και θα πρέπει οι χώρες μέλη να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν, να λαμβάνουν, να του επιστρέφονται τα έξοδα για τις ε, εκθέσεις και ε, μέχρι στιγμής 5%. Επίσης τα μέσα της Κομισιόν θα πρέπει να αυξηθούν, τα κονδύλια, εφόσον η πληρωμή γίνεται ευθύ εξ αρχής και κατά 100%. Και αυτή είναι μια δημορφία του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή ότι είναι δυνατόν ευθύ εξ αρχής να πάρει κανείς το 100% των χρημάτων. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί σε περιπτώσει όπου γίνεται κάτι τέτοιο και γινόταν αυτό στο παρελθόν να μπορεί να διευρυνθεί η δυνατότητα ελέγχου εκ μέρου τη Επιτροπή. Πρόκειται δηλαδή για ένα στοιχείο το οποίο δεν το γνωρίζουμε από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, σφάλματα τα οποία διαπιστώνονται θα πρέπει να διορθώνονται άμεσα μέσω συμψηφίσμου και εάν βλάπτονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις. Αυτές οι τροπολογίες 10 και 11 αυτό λένε και πέραν τούτου θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Δηλαδή ε, το εργαλείο μέσω των εργαζόμενων που υποφελούνται από αυτό θα πρέπει να έχει πραγματικά μια χρησιμότητα και να μην αντικαθιστά κατ' ουσία κάποιες ε, λειτουργίες του δημοσίου. Γιατί μέχρι τώρα αυτά ήταν χρήματα που θα δίδανταν από, το εκάστοτε, ε, από την εκάστοτε χώρα μέλος και τώρα δίδονται από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ε, τα κονδύλια αυτά δεν ε, περιλαμβάνονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει μια εντονότερη συμμετοχή του ελεγκτικού συνεδρίου. Η τελευταία τροπολογία υπαριθμών 12 αναφέρεται στις κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτό είναι ένα όμως μόνιμο θέμα μεταξύ, συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα και θα ήθελα να χαιρετήσω τον ζάν Φρανσουά Λεπράν από την Επιτροπή. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε κύριε Λεμπράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις έχοντας διαβάσει και ακούσει ε, τα σχολεία για τροπολογίες του εισηγητή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι θα ήταν χρήσιμο ίσως να προσεγγίσουμε διαφορετικά την ιστορική διαδρομή αυτού του ταμείου. Ο στόχος του δεν είναι να καταστήσει πιο δημοφιλές και με συμβολικό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος ήταν να χρησιμεύσει αυτό το ταμείο για να ε, ε, δείξουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μετά από αναδιαρθρώσεις, μετά από μαζικές απολύσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι είναι θετική η παγκοσμιοποίηση για τους περισσότερους, αλλά ε, ορισμένες φορές έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμο να δείχνουμε αλληλεγγύη με τους εργαζομένους που δυστυχώς πλήττονται από αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μόνο μεγάλες κλίμακας αναδιαρθρώσεις δυστυχώς και παρεμβαίνουμε ούτως ώστε ένας απολυμένος να έχει τη δυνατότητα να ξαναβρει δουλειά βάσει ε, μέτρων ενεργητικής πολιτικής, έτσι ονομάζονται, στην αγορά εργασίας έχουν ήδη επωφεληθεί από το ταμείο αυτό πολλοί εργαζόμενοι και δεν είναι συμβολική η αξία του. Ήταν μια ουσιαστικότατη βοήθεια που προσέφερε για λόγους αλληλεγγύης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πιστεύω και ευχαριστώ τον εισηγητή για το άνοιγμα που κάνουμε στον τομέα της γεωργίας, διότι μέχρι του δηλαδή στην τωρινή περίοδο προγραμματισμού, η γεωργία και πιο συγκεκριμένα η μικρή γεωργοί, ανεξάρτητοι επαγγελματίες που έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις, δεν καλύπτονται. Με αυτό το νέο άνοιγμα του Ταμείου κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να επικρατήσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Ε, ως προς την ε, οικονομική κρίση, το 2009, το που εκδηλώθηκε η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, παρατάθηκε το πεδίο εφαρμογή ε, του. Επεκτάθηκε, συγγνώμη, το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για να καλύψει και την κρίση. Σταμάτησε φέτος ε, αυτή η νέα προσέγγιση. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει γι' αυτό επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που ακόμη υπάρχει ε, το Κοινοβούλιο είχε εξάλλου εγκρίνει αυτή την εξαίρεση. Τώρα, στη νέα περίοδο προγραμματισμού προβλέπουμε το κριτήριο της απροσδόκητης κρίσης για να μπορέσουμε να καλύψουμε διάφορα αίτια της κρίσης, οικονομικής κρίσης, ε, κρίσης ε, στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε κρίση που ενδέχεται ε, με μόνιμο τρόπο να επηρεάσει την εθνική παραγωγή. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν το Κοινοβούλιο που μας υποστηρίζει διότι ξέρετε ότι στις συζητήσεις στο Συμβούλιο δεν υπάρχει τέτοια προθυμία. Ε, αναφερθήκατε στις ενιαίες πληρωμές, πληρωμές 100%. Για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτή τη λύση. Εφόσον δεν εντασσόμεθα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, οποιοδήποτε αίτημα ε, στήριξης παρατείνεται χρονικά Δηλαδή πρέπει να καταμετρηθούν οι απολύσεις σε εθνικό επίπεδο, να προετοιμαστεί το πρόγραμμα. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύσει και να αξιολογήσει το εθνικό πρόγραμμα για να διαπιστώσει αν υπάρχει συμμόρφωση με τα διάφορα κριτήρια που προβλέπονται στη, στον κανονισμό και τέλος χρειάζεται συζήτηση στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο κτλ. Συχνά η διάρκεια ανέρχεται σε ένα χρόνο, ανάμεσα δηλαδή στη χρονική στιγμή της απόλυσης και την εκταμείευση της πληρωμής. Δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν ήδη επενδύσει ένα τμήμα της ενίσχυσης. Ε, θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε μια πιο μαζική παρέμβαση, κυρίως γιατί σε πολλά κράτη-μέλη περιμένουν το πράσινο φως από τις ε, δημοσιονομικές αρχές της Ένωσης για να αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Χρειάζεται επίσπευση λοιπόν για να επωφεληθούν οι ούχοι ε, και πέρα από αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση είχαμε και περιστατικά ε, ανάκτησης ποσών. Τα κριτήρια είναι σαφέστατα. Αυτό αποδεικνύεται από το εξής. Κανένα αίτημα παρέμβαση δεν έχει απορριφθεί ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στο Σύμβουλιο. Αν κάνουμε τώρα μία σύγκριση με το Ταμείο Αλληλεγγύης για τις φυσικές καταστροφές, διαπιστώνεται πολύ μεγάλες διαφορές που μπορούν να αποδοθούν στην σειρά κριτηρίων που προβλέπει ο βασικός κανονισμός. Σε σχέση με τις κυρώσεις τώρα που προτείνεται, μπορεί κανείς να προτείνει κυρώσεις, αλλά η εμπειρία μας μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν υπήρξε λόγος μετά από τους διαδοχικούς ελέγχους και αξιολογήσεις να κάνουμε κάτι τέτοιο και το διαπιστώνουμε συχνά στη μονάδα ελέγχων. Έχουμε ανάκτηση ποσών ενίοτε, αλλά δεν υπήρξε δόλο σε καμία περίπτωση. Τώρα αναλύουμε το IGF και ίσως αυτό καλύπτει τις, τους προβληματισμούς σας για την εμπλοκή του ελεγκτικού συνεδρίου στην ανάλυση κατάστασης και τη χρήση αυτού του ταμείου. Τώρα, σε σχέση με τις εθνικές πρωτοβουλίες για το θέμα που αποκαλούμε τεχνική αρρωγή και που έχετε τοποθετήσει στο 5%. Βάσει των στοιχείων μας, ο μέσος όρος μέχρι στιγμής είναι 4%. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπήρξε υπέρβαση ε, αλλά ήταν ε, αιτιολογημένε από τι εθνικέ αρχέ. Σε παράδειγμα, σε περίπτωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γιατί ξέρετε ότι και σε τομεακό επίπεδο μπορούμε να παρέμβουμε. το ότι μπορούμε να ε, καταγράψουμε όλε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τους εργαζομένους ε, που είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες ε, γεωγραφικές περιοχές. Αυτό επιφέρει μεγαλύτερο κόστος. Είναι βεβαίω αυτονόητο σε ορισμένε περιπτώσει, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να τεκμηριωθεί και άρα χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα κριτήρια τώρα για να περάσουμε για το ποσοστό ε, συγχρηματοδότηση από το 50% στο 65%. Χρειάζεται η ισορροπία ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι σαφέστατα κριτήρια, μεγαλύτερη πειθαρχία και αυτό καλύπτεται από τον κανονισμό για τον αριθμό των απολύσεων, για το είδος ε, των γεωγραφικών περιοχών. Υπάρχει μια ε, σειρά άκαμπτων, αν θέλετε, κριτηρίων, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και μια ευελιξία, ώστε η παρέμβασή μας να είναι η πλέον πρόσφορη στις περιπτώσεις που ε, μας προτείνει κάθε κράτος μέλος. Ε, τα κριτήρια για να περάσει κανείς από το 50% στο 65% είναι σαφώς προσδιορισμένα εκ των προτέρων. Χρειάζεται πάντως σωστή ισορροπία ανάμεσα στα αυστηρά συγκεκριμένα κριτήρια και την ευελιξία που χρειαζόμαστε για την πρακτική εφαρμογή. Αυτά που λέμε στην έκθεση για τον αριθμό των εργαζομένων που μπόρεσαν μέσα σε ένα χρόνο να βρουν μια σταθερή θέση εργασίας και άλλα τέτοια στοιχεία μπορούν όντως να μας φανούν χρήσιμα. Στο Συμβούλιο ήθελα να σας ενημερώσω ότι συζητήσαμε ε, για τον ορισμό τη σταθερή θέση απασχόληση. Καταλαβαίνω ότι κάθε νέο στοιχείο μπορεί να οδηγήσει σε ατέρμονε συζητήσει. Ειδού κάποια στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν, ελπίζω, το προβληματισμό και το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέμπρα. Υπάρχουν ερωτήσεις; Θέλει να παρέμβει ο εισηγητής, θέλει να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ, κύριε Χάτζη Μαρκάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αισιοδοξία που δείχνει η Επιτροπή. Δηλαδή, ε, το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, το πολύ, 100, στην καλύτερη περίπτωση 133 εκατομμύρια είναι ενδεικτικό. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν απορροφώνουν τα ποσά, τα 500 εκατομμύρια που έχουμε ετσίως. Δεν θα πρέπει να πατώμεθα. Όταν ε, θέλουμε απλώς να κάνουμε χειρή την παρουσία μας, αλλά δεν γίνεται αντιληπτή, νομίζω ότι πρόκειται μόνο για κονδύλια ε, τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούνται. Ε, αυτά έτσι κι αλλιώς είναι απομεινάρια από άλλα ταμεία όπως σας είπα. Αλλά χαίρομαι που ψάχνετε κάποιους τρόπους για να αντιδράσετε με ευελιξία και ταχύτητα. Ε, χαίρομαι που συμπεριλαμβάνονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μαζί με τους ε, γεωργούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη νομίζω ότι, δεν θα, ε, ότι θα πρέπει να έχετε πιο αυστηρά και πιο ξεκάθαρα κριτήρια. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Όχι, ο κύριος Λεμπρέν θέλει να δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυσμόνησα να δώσω μια απάντηση όσον αφορά το ποσό που ανέφερε ο εισηγητή στα ποσά. Ε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πρόκειται σαφώς περί ενός ταμείου που είναι εκτός του προϋπολογισμού που έχει δυνατότητα η μέγιστη κινητοποίησης 500 ε, εκατομμυρίων. Το ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτό το ταμείο, αυτού του πόρου, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα για τα στοιχεία που βρίσκονται εντό του δημοσιονομικού πλαισίου. Το ότι αυτό είναι συμπληρωματικό ταμείο συμπληρώνει τι δράσει που μπορούν να ασκήσουν οι επιχειρήσει, οι δημόσιε αρχέ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα είχα την τάση να πω ότι αν σε όλες τις χώρες είχαμε συστήματα που θα επέτρεπα να διαχειριστούμε την αναδιάρθρωση με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουμε. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό. Ο στόχο όσον αφορά όμω την κοινωνική πολιτική για ένα τέτοιο ταμείο είναι η χρήση 0 ευρώ. Όσο λιγότερο το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερο θα έλεγα, καλύτερη είναι η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεμπρά. Με τη συμπλήρωση αυτή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης μας σήμερα. Προπολογισμό 2013. Πρόκειται για την εντολή για τον τριμερή διάλογο και θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή, τον Κρίστοφερ Φιέλνερ και να τον παρακαλέσω να μας κάνει την παρουσίαση. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος, παραδοσιακά είναι κάτι που ακολουθεί σαν λογική συνεπαγωγή όταν είναι κανείς ε, εισηγητής για την απαλλαγή κάνει και αυτό το θέμα. Συγγνωμοδότησή μου προσπάθησα να εστιαστώ επί ενός θέματος ουσιαστικά. Και θα αναφερθώ και στο ψήφισμα της απαλλαγής επ' αυτού. οι εκρεμείς υποχρεώσεις του προϋπολογισμού. Βλέπουμε ότι βασικά απορρέουν από πολιετή προγράμματα, κυρίως συνοχή. Βλέπουμε και σημειώνουμε αύξηση. Σημαντική. Το 2010 αύξηση περίπου 10% και ξέρουμε ότι παρόλο που κατά κάποιο τρόπο υπάρχει διακύμανση κατά την προγραμματική περίοδο και πάλι σημαίνει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα κυρίως εντός της οικονομικής κρίσης. Και αυτές οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις ίσως δείχνουν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απορρόφηση των ποσών που τους διατίθενται. Όταν συζητούμε τον προϋπολογισμό, για το 2013 το σχέδιο προϋπολογισμού πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη δύνανται να απορροφήσουν τους πόρους που τους διατίθενται. Και γι' αυτό χρειάζεται διεξοδική ανάλυση στον προϋπολογισμό του 2013 και στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο εξίσου σημαντικό στο τέλος, αυτό που αναφέρω. Συζητείται εκτενώς το θέμα των ιδίων πόρων. Τι είδους ιδίους πόρους διαθέτουμε, Φαίνεται να εφευρίσκουμε κάθε εβδομάδα νέους ίδιους πόρους. Και όποιο εισόδημα και αν επιλέξει κανείς, έχει διαφορετική επίδραση στην οικονομία. Πρέπει να δούμε τα διάφορα είδη λοιπόν συλλογή εισοδήματο και πώς γίνεται η επιλογή της πηγής. evaluated revenue collection for the European Union. Uh, as I said, mainly it's a call on the negotiation. Οι διαπραγματευόμενοι πρέπει να δουν το θέμα των εκκρεμών υποχρεώσεων. Πρέπει να εξεταστεί, κυρίως αν τα κράτη-μέλη έχουν δυσκολία όσον αφορά την απορρόφηση των χρημάτων. Αυτά. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Όσον αφορά τις εμπειρίες για την απορρόφηση, ποσοστά απορρόφησης και δυνατότητες απορρόφησης, υπέβαλα έκθεση στο Κοινοβούλιο για συνοχή, ταμεία συνοχής και τα τα ταμεία. Και το θέμα απορρόφησης που θέσατε είναι σημαντικό Στηρίζω αυτή την άποψη. Η κυρία Τζένιφερ Μπράουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας πάρει το λόγο τώρα. Έχετε το λόγο κυρία Μπράουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αύριο. Και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι πάει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού άρα δεν θα αναφερθώ σήμερα σε λεπτομέρειες, διότι μένει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις εκκρεμούσες ε, υποχρεώσεις ή τα ραλ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις των ραλ που προέκυψαν ε, το 2011 και έφτασαν τα 207 δισεκατομμύρια. Να υπενθυμίσουμε, τα, τα υπόλοιπα προς ακαθάριση ραλ είναι φυσική συνέπεια διαφοροποιημένων δεσμεύσεων και πληρωμών του προπολογισμού και μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια θα είναι η αιτήσια αύξηση των υπολείπων προς εκαθάριση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληρωμές και να τι αφαιρέσουμε από τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Άλλα στοιχεία παίζουν ρόλο βέβαια. Κανονικό είναι, όπως είπε ο συγητής, ότι σε διάφορα σημεία της προγραμματικής περίοδου τα υπόλοιπα προς εκαθάριση διακυμαίνονται. Περισσότερε αναλήψει υποχρεώσεων στην αρχή τη περίοδου και περισσότερε πληρωμέ προ το τέλο έχουμε. Οπότε το ράλι είναι υψηλό τώρα, αλλά θα καλυφθεί τελικά από τις τελικές πληρωμές και την εκτέλεση υποχρεώσεων στο τέλος της περίοδου. Περίπου 50% των κατεκαθάρισεων ποσών προέρχεται από το 1β και με, πηγαίνοντας από το 1-2 προς το 1-3 λόγω οικονομικής κρίσεως αναπτύχθηκε περισσότερο το ΡΑΛ. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των υπολείπων σε καθάριση ποικιλοτρόπω. Να μειώσουμε τι αναλήψει νέων υποχρεώσεων στον προπολογισμό, δυσκολότατο, σε πολιτή προγραμματισμό. Δεύτερη προσέγγιση, αύξηση του επίπεδου των πληρωμών. Αλλά οι πρόσφατες διαδικασίε του προπολογισμού έδειξαν πόσο πολιτικός δύσκολο είναι αυτό και πόσα αντιστάσει υπάρχουν στο Συμβούλιο για κάτι τέτοιο. Άλλη δυνατότητα, να καταργηθούν υποχρεώσεις αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε. εν συν 3 παραδείγματος χάρη. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα των υπολείπων προς εκαθάριση, η ΡΑΛ, και όπως είπε ο συγητή, είναι πολύ σημαντικό στα, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του προπολογισμού. Κρίσιμο στοιχείο είναι το εξή. Στις διαπραγματεύσεις καταφέρουμε να γερώσουμε χάσματα μεταξύ αναλήψη υποχρεώσεων και εκτελές πληρωμών. Και στι τελευταίε δύο διαδικασίε του προπολογισμού είδαμε ότι αυτό είναι δύσκολο. Η ανάληψη υποχρεώσεων αυξανόταν σημαντικά και οι πληρωμές έμεναν αρκετά χαμηλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση. Πρόκειται για 207 δις στο τέλος του 2010 ή του 11. Του 11. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπράουν και τώρα ο εισηγητής έχει το λόγο. Ε, πάρα πολλά χρήματα είναι επικίνδυνα τα πράγματα με τόσο μεγάλα νούμερα. Είναι πραγματικά φοβιστικά. Ε, με εξέπλεξαν δύο πράγματα και ίσως είναι τα απομεινάρια από την απαλλαγή. Θα ήθελα να αναφέρω όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε θεωρώ πιο προσεκτικά στην Επιτροπή στο μέλλον. Καταρχήν, και πράγματι το έχουμε κάνει αυτό σε διάφορες περιπτώσεις, έχουμε αυξήσει το επίπεδο πληρωμών, ε, συνεπία της χρηματοπιστωτικής κρίσης κλπ. νομίζω ότι αν αυξήσουμε το επίπεδο των πληρωμών και επιταχύνουμε το 1 συν 2 κλπ, ε, εδώ υπάρχει το ζήτημα του περιθωρίου σφαλμάτων. Εάν αλλάξουμε τους κανόνες, ε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω κάποιες ανησυχίες και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε κατά νου στην Επιτροπή. Και τέλος, κάτι ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχω, ε, έχω τους αριθμούς ε, όσον αφορά την απαλλαγή, αλλά δεν είχα τον καιρό να τα κοιτάξω. Όσον αφορά τα ραλ, το ζήτημα είναι ποιες χώρες αφορά και πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί πάντοτε ακούμε ότι πρέπει να κάνουμε το ένα ή το άλλο ε, συνεπία της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αλλά πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο ότι έχουμε τα περισσότερα ραλ τα οποία κατανέμονται στις χώρες που αντιμετωπίζουν πιο έντονη χρηματοπιστωτική κρίση. Νομίζω θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα των υπολείπων προς εκαθάριση των ε, ραλ. Ε, να δούμε τι γίνεται στις 17 χώρες και τα προγράμματά τους και να θεωρήσουμε αν πράγματι τα προβλήματα είναι εκεί που θεωρούμε ότι βρίσκονται ή θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποιο άλλου είδους διαθωτικά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ Κρίστοφερ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι σημαντικό το θέμα αυτό το οποίο δείχνει η θα πρεπει να εντοπισουμε καποιο αλλο ειδους διαφορετικα προβληματα ευχαριστουμε πολυ κριστοφερ νομιζω οτι πραγματικα ειναι σημαντικο το θεμα αυτο το οποιο δειχνει η εκθεση για τις ε, δυνατότητες ε, απορρόφησης των ε, ποσών. Ε, για παράδειγμα στα περιφερειακά και διευθυντικά ταμεία. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η Εσθονία που έχει πολύ ψηλά ποσοστά απορρόφησης και ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που έχουν χαμηλά ποσοστά απορρόφησης. Αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο, θα πρέπει να το δούμε πιο πολύ εκ του σύνεγγες, να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι γιατί είναι πολύ εύκολο να βλέπει κανείς μόνο τα αποστάσει χρηματοδότησης. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποια άλλα εμπόδια ε, σε σχέση για παράδειγμα τις δομές λήψης αποφάσεων κλπ. Ε, μπορούμε να έχουμε από την Επιτροπή κυρία Μπράουν μια απάντηση όσον αφορά την ανάπτυξη των ταμείων. Μπορείτε δηλαδή να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με τα ΡΑΛ αν βρίσκονται κυρίως σε συγκεκριμένες ε, γραμμές του προπολογισμού ή όχι. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Τα, το βασικό τμήμα των ΡΑΛ, περίπου το 50% σχετίζεται με, το, με την κατηγορία 1β, με τις ε, δομικές ε, διαθροντικές δράσεις, σε σύνδεση με την ανάπτυξη της υπαίθρου που έχει μια παρόμοια δομή και αν συμπεριλάβουμε και αυτό θα φτάσουμε στα δύο τρίτα των ραλ. Με όρους απορρόφησης, ωστόσο, υπάρχουν ότι υπάρχει μια επιτάχυνση και αυτό συνέβη ξεκάθαρα στα τέλη του 2011 όπου υπήρξε πραγματικά μια πλημμυρίδα ετοιμάτων πληρωμών από τις χώρες μέλη ε, ε, και έμειναν 11 εκατομμύρια ε, τα οποία δεν είχαν πληρωθεί. Ε, σε προβλήμα του προπολισμού του 2011. Αλλά υπάρχουν κάποια παραδείγματα όπου υπάρχει μια τέτοιου είδου επίσπευση. Ιδιαίτερως όσον αφορά ε, την εφαρμογή των κανόνων N 1 ή N 2 που κάποιοι, κάποιες χώρες έκαναν πιο πολλές προσπάθειες να επιταχύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπράουν. Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και την γραμματεία γιατί πραγματικά είχαμε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Σήμερα είχαμε την ακρόαση και την οποία προτίμασε πολύ καλά ο κύριος Νέρλιχ. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν επίσης στην επιτυχημένη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. Ευχαριστούμε και τους ερμηνείς.